Σας παρακαλώ να καθίσετε και ε, όσοι είστε μέλη να έχετε μαζί σας τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Λοιπόν, για να δούμε, είναι εδώ και ο συντονιστής της ομάδας μου. θυμάμαι 40 χρόνια πριν, όταν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λίβερπουλ, ε, πάντα αργούσε αυτό ο ένα από τον οποίο εξαρτιόταν αν θα περάσει όχι, από την ψήφο του, αν θα περάσει ή όχι ένα θέμα. Και ήταν Πάντα αργοπορημένος, πάντα. Εν πάση περιπτώσει, τα δικά μας τώρα. Πρώτο, σύσταση επί της αποφάσεως ε, του Συμβουλίου για βιώσιμη εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Γκάμπια. Ε, η συγγετρία του Κοινοβουλίου προτείνει να ψηφίσουμε υπέρ, άρα να ψηφίσουμε. Ωραία, ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συστάσεως αυτής. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, ε, μία ψήφος κατά, 6 αποφιές. Δεύτερο θέμα και δεύτερη ψηφοφορία λοιπόν. Αυτή αφορά την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Αλίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ο εισηγητής είναι υπέρ για μία ακόμα φορά. Απαιτείται πλειοψηφία ψήφων στην Επιτροπή μας, δηλαδή 15 τουλάχιστον, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. και εγκρίνεται με 20 θετικές ψήφους, 6 αρνητικές, 2 αποχές. Ωραία, τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. So we now proceed with the uh, hearing. Επομένως τώρα θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου της Αλίας. Έχουμε βεβαίως πρώτα απ' όλα και υπόψη μας ένα προσχέδιο κανονισμού από την Κομισιόν. Ε, αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Παλιότεροι βουλευτές θα θυμούνται ότι έχει ξανασυζητήσει το θέμα ε, επανειλημμένα και τώρα θα το ε, συστήσουμε και στα νέα μέλη. Καλωσορίζω τους ομιλητές μας. Ε, τους υπενθυμίζω ότι θα τους παρακαλούσαμε να μην ξεπεράσουν τον χρόνο που τους έχει δοθεί, δηλαδή τα 10 λεπτά. Και θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στην Κομισιόν για μια σύντομη εισαγωγή. Παρακαλώ Κομισιόν, η κυρία Αρένα νομίζω θα μιλήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα βγάζετε τα χαρτιά σας κυρία Αρένα, σας περιμένουμε. Θέλετε όμως να μας ε, κάνετε μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τον νέο κανονισμό για τον έλεγχο της αλληλείας. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ε, μέλη της ε, Επιτροπής σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας. Η Κομισιόν ήδη είχε σε άλλες περιπτώσεις την ευκαιρία ε, να παρουσιάσει ενδελεχώς την πρόταση ε, σχετικά με ένα ε, νέο έλεγχο, σύστημα ελέγχου. Αυτό έγινε εδώ στην Επιτροπή Αλληλείας τον Ιούλιο του 2019. Θα... Ήθελα να πω ότι όπως γνωρίζετε η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει φιλόδοξους στόχους οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μονάχα εάν όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της διαθέτει ε, σύστημα ε, έλεγχου αποτελεσματικό και σύγχρονο. Μπορεί κανείς να έχει όσα μέτρα, όσες προβλέψεις, όσα νομοθετικά κείμενα, αλλά εάν αυτά και τα μέτρα τα οποία σε αυτά περιλαμβάνονται δεν ε, εφαρμόζονται και δεν υπάρχει έλεγχος εφαρμογής, τότε δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Άρα ο έλεγχος κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να θεωρηθεί η σπονδυλική στήλη του συστήματος. Αναμφίβολα ε, το πλαίσιο ελέγχου της αλληλείας ε, που ήδη ε, ισχύει και υιοθετήθηκε πριν από 10 χρόνια αποτέλεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προόδου και οπωσδήποτε η πλήρης εφαρμογή ε, του υφισταμένου συστήματος παραμένει προτεραιότητα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίστηκε γενικώ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων ότι το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προετοιμαστεί έτσι ώστε να είναι σε στην να αντιμετωπίσει τις του μέλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν έγινε δεκτή η πρόταση αναθεωρημένης ε, πρότασης για τον έλεγχο της ε, αλίας που αφορούσε και τον έλεγχο αυτόν καθεαυτό και τον ε, κανονισμό χρηματοδότησης της αλίας καθώς επίσης και το κείμενο για την παράνομη άναρχη αλία. προτάθηκαν με κάποιες λύσεις από την Κομισιόν ε, για προβλήματα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ε, ότι υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα ε, η πολιτισμική συμμόρφωση δεν γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, και δεν εφαρμόζονται καλά οι κυρώσεις, ε, δεν δίνονται οι απαραίτητες, ε, τα απαραίτητα points σε περιπτώσεις παραβιάσεων και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά την έννοια ότι προκαλεί μεγάλη στρέβλωση Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει την απλοποίηση των διατάξεων και την εναρμόνισή τους μέσω ε, κοινής, κοινού καταλόγου σημαντικών παραβάσεων που θα ισχύουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνει επίσης σταθερά κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνεται η σοβαρότητα της παράβασης καθώς επίσης καθορίζονται και μέγιστα όρια κύρωσης επί τη βάση ε, της, ε, του αλλιεύματος στην συγκεκριμένη παράβαση. Και με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί ο βαθμός συμμόρφωσης, ε, καθώς επίσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί η βιωσιμότητα σε σχέση με τους ε, πόρους. Δεύτερο πρόβλημα το οποίο ταυτοποιήθηκε είναι η επιτήρηση της αλλιευτικής δραστηριότητας ε, και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή. Όταν συζητούμε, όταν μιλούμε για έλεγχο, ε, θέλουμε να ξέρουμε ό,τι συμβαίνει. Ποιος ψαρεύει, τι, πού και πόσο. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας έτσι ώστε ε, ε, να ε, ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, όσον αφορά τις ποσότητες κλπ. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν επίσης δυνατότητα στους επιστήμονες να καθορίσουν την κατάσταση των αποθεμάτων έτσι ώστε με τη σειρά τους να δώσουν στοιχεία στους διαχειριστές που θα ορίσουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Ε, ε, στην παρούσα κατάσταση υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυνατότητες πολλές δυνατότητες ε, για μία αναφορά των ε, στοιχείων ε, προς Δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε τις παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα στο βαθμό που θα θέλαμε και επομένως να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης ξέρουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα όσον αφορά την ερασιτεχνική αλληλεία και για, την, για τα πολύ μικρή κλίμακος εμπορικά σκάφη επίσης δεν έχουμε σχεδόν καθόλου πληροφορίες. Όλα αυτά τα στοιχεία παρεμποδίζουν την ε, λήψη ασφαλών αποφάσεων από τους διαχειριστές. Επομένως, η Κομισιόν προτείνει πλήρη ψηφιοποίηση των ε, δεδομένων ε, της αλίας, ε, να ξεχάσουμε τα συστήματα που βασίζονται σε χρήση χάρτινων υποδομών και επίσης μέσω της ψηφιοποίησης να έχουν ε, όλα τα σκάφη ε, ε, συστήματα εντοπισμού και υπολογισμού των αλλιευμάτων ανεξαρτήτως του μήκους τους και μέσω χρήσης πολύ απλών συσκευών, όπως ας πούμε τα smartphones, να απλουστευτεί η διαδικασία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα τρία τέταρτα των νέων σκαφών είναι κάτω από 14 μέτρα ε, και επομένως για αυτά ε, βάσει του παλαιού συστήματος δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα εντοπισμού και ελέγχου. Να σας υπενθυμίσω επίσης ε, ότι το λεγόμενο green box είναι ένα σύστημα ε, το οποίο αφορά τον εντοπισμό όλων των σκαφών και απεδείχθη ένα σύστημα πολύ απλό και εύχριστο. Επίσης, επομένως, εισάγονται ε, κάποιοι κανόνες και άλλοι ενδυναμώνονται όσον αφορά την αριστε... Ε, ερασιτεχνική αλληλεία, γιατί υπάρχει και ένα σκέλος εμπορικής αλληλείας και εδώ. Το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ευθυγράμμιση με την κοινή αλληλευτική πολιτική το ε, ε, ισχύον σύστημα ελέγχου, αυτό δηλαδή του 2009, δεν μπορούσε να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το πι, ε, κυρίως όσον αφορά το θέμα των εκφορτώσεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αντιμετωπίζεται με τη νέα πρόταση της Κομισιόν. Προτείνεται λοιπόν να μειωθεί αυτό αυτή η υφιστάμενη διαφορά μέσω ε, ενός συστήματος διαρκούς επιτήρησης των δραστηριοτήτων στην θάλασσα μέσω τηλεεπιτήρησης. Αυτά τα εργαλεία ηλεκτρονικής εξαποστάσεως ε, επιτήρησης ε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα υψηλό ποσοστό των πλοίων, των σκαφών, σύμφωνα με τις μελέτες ε, που έχουμε κάνει. Με τις τρεις προτάσεις αυτές που ανέφερα ή τα τρία στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως, οπωσδήποτε μπορεί να ε, έχουμε ε, πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και όσον αφορά την επιτήρηση των σκαφών, όσον αφορά την εκφόρτωση απλών ή μεταποιημένων προϊόντων, ε, ε, προτείνουμε ένα σύστημα λιγότερο περίπλοκο όσον αφορά ε, την, την, τον έλεγχο και την επιτήρηση της ισχύω των μηχανών ε, και ε, ε, να τελειώσει πλέον αυτό το σύστημα των πολλαπών εξαιρέσεων το οποίο ισχύει σήμερα. Η Κομισιόν επίσης προβλέπει κάποιες νέες διατάξεις όσον αφορά την ΕΦΚΑ, την υπηρεσία ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλίας στην οποία θα δοθούν κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες όσον αφορά τις ε, διεθνείς δραστηριότητες. Αυτά ε, ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι σας έκανα μια ε, σύνοψη της πρότασης και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις αργότερα κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ε, Κομισιόν. Μας βάλατε λοιπόν λίγο στο κλίμα. Θέλουμε όλοι βιώσιμη αλληλεία, θέλουμε όλοι να σταματήσει ε, ο αποδεκατισμός των ε, αποθεμάτων, θέλουμε ε, να έχουμε ένα, έχουμε ένα μέλλον ευημερία και επιτυχίας για την αλλιευτική μας βιομηχανία και τον αλλιευτικό κλάδο. Ε, βεβαίως, ε, και η Κομισιόν το είπε, ε, πολλά ε, πολλά εύματα δεν καταγράφονται ε, και θα πρέπει να δούμε σε αυτές τις παραβάσεις τι είδους κυρώσεις και πώς μπορούν να ευθυγραμμιστούν αυτές οι κυρώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε εμπειρογνώμονες ε, που περιμένουμε να τους ακούσουμε με ανυπομονησία. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πασκάλ Σαβουρέ, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλληλείας. Εύκα, κύριε Σαβουρέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα σε αυτή την ακρόση. Τα δέκα λεπτά που μου δώσατε θα τα αφιερώσω στην παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποιες από τις ε, επιθεωρήσεις και παρακολουθήσεις που κάνουμε με αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που βρίσκονται επί των σκαφών. Γιατί θέλω να σας παρουσιάσω αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την απαγόρευση απόρριψης, discard ban στα αγγλικά, και τις δυνατότητες ε, απορρίψεων που συνεχίζουν να επιτρέπονται και να είναι συμβατές με την ε, βασική, αν θέλετε, ρύθμιση και τον κανονισμό που διέπει την κοινή πολιτική. Πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως όμως με αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι το κοινό σήμερα γνωρίζει ότι υπάρχει το σύστημα της τηλεόρασης ε, κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται επί των σκαφών και που παρακολουθεί με έναν μεγάλο αριθμό αισθητήρων την δραστηριότητα, ακριβώς τι συμβαίνει με όλο τον εξοπλισμό, τα βίντζια, την ένταση των ε, ηλεκτρικών συστημάτων, τη θερμοκρασία στα αμπάρια, τα ανοίγματα των αμπαριών, τις πόρτες, τις δεξαμενές, καθώς και την ε, λεγόμενη δραστηριότητα του Power Block, δηλαδή στα ελληνικά οι τροχαλίες, οι αντλίες, αλλά και οι βαλβίδες ε, και οι ε, πόρτες των αμπαριών και των κάδων. Υπάρχει μια ολόκληρη λοιπόν σειρά μηχανημάτων εξοπλισμών που θα πρέπει να παρακολουθούνται εξ αποστάσεων και αυτή η μελέτη Βεβαίως, αν σας ενδιαφέρει σε όλες τις λεπτομέρειες, υπάρχει στην, στον ιστότοπο της υπηρεσίας ελέγχου της αλίας για όποιον θέλει περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως, καταρχήν πρέπει να υπάρχει η συμμόρφωση του επικεφαλής του σκάφους, του ιδιοκτήτη, αλλά και κυρίως όλων των χειριστών και των αλλιέων. Όσον αφορά την, ε, τα επιτρεπόμενα όρια απορρίψεων, αυτά θα πρέπει να είναι γνωστά και να δούμε ποιες είναι οι διατάξεις αυτές οι οποίες ουσιαστικά δικαιολογούν και ερμηνεύουν αυτόν τον ε, έλεγχο, τον επιπλέον έλεγχο δηλαδή που διεκπεραιώνεται με ηλεκτρονικά συστήματα πάνω στα σκάφη. Υπάρχουν κάποιες από τις διατάξεις της κοινή αλλιευτικής πολιτικής που ουσιαστικά αναγνωρίζουν ότι κάποιες παρεκκλήσεις από την ε, πλήρη απόρρι... Ε, απαγόρευση απορρίψεων υπάρχουν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κανονισμός στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής προβλέπει ότι χρειάζεται παρακολούθηση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αλλιεύματα και αποθέματα τα οποία υπόκεινται στα όρια είτε όταν υπάρχει θέμα μεγέθους για αποθέματα παραδείγματος χάρη τα οποία έχουν ε, ε, αλλιευθεί και τα οποία βρίσκονται σε πάρα πολύ ε, μικρά μεγέθη. Για αυτές τις περιπτώσεις αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται αμέσως. Βεβαίως, η απόρριψη δεν είναι απαραίτητα παραβίαση του κανονισμού. Και εδώ θα αναφερθώ στο άρθρο 15, γιατί όταν υπάρχει παραβίαση όσον αφορά την εκ, μη εκφόρτωση κάποιων ε, αποθεμάτων που υπόκεινται στα όρια, το πρωτόκολλο παρακολούθησης και ελέγχου, το οποίο ουσιαστικά βασίζεται σε έλεγχο, επιτήρηση, αλλά εδώ θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες παρακολούθησης. Στο άρθρο 73 του κανονισμού που αφορά τον έλεγχο, προβλέπεται η υλοποίηση αυτής της έννοιας της παρακολούθησης. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει χώρος επιτόπου στα αλλιευτικά σκάφη. Επίσης, η παρακολούθηση από κάποιον ε, υπάλληλο δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει απαραίτητος χώρος στα αλλιευτικά σκάφη και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται 24 ώρες το 24 ώρο, αυτό είναι αδύνατο. Γι' αυτό και θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις από μέρους των πληρωμάτων των αλλιευτικών σκαφών, να λειτουργούν τα συστήματα ε, παρακολούθησης και βεβαίως όσον αφορά τις απορρίψεις να απορρίπτονται στην θάλασσα μόνο τα είδη και τα αποθέματα αυτά για τα οποία υπάρχει άδεια. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής εξαποστάσεων παρακολούθησης, οι οποίες προτείνουμε να εγκατασταθούν στα αλληλευτικά σκάφη, θα κάνουν την υπόλοιπη συμπληρωματική παρακολούθηση. Ποια είναι η δική μας άποψη, η άποψη της δικής μας υπηρεσίας επ' αυτού. Καταρχήν θεωρούμε ότι ο τομέας της αλίας δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει πλήρως ε, τις ε, υποχρεώσεις να συμμορφωθεί με τους κανόνες που ορίζουν την υποχρέωση εκφόρτωσης. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί. Το σύστημα της μέχρι τώρα παρακολούθησης και ελέγχου ουσιαστικά βασίζεται σε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες ουσιαστικά μπορεί να ληφθούν παρουσία του επιθεωρητή, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι η ίδια συμπεριφορά συνεχίζεται και μετά την αποχώρηση του ελεγκτή, του επιθεωρητή. Τα ίδια σκάφη λοιπόν και τα ίδια αλλιεύματα με κάμερες και χωρίς κάμερες δεν έχουν καθόλου τα ίδια αποτελέσματα. Είδαμε δηλαδή ότι πολλές φορές ε, οι δηλώσεις που κάνουν ε, οι αλλοίς ουσιαστικά δεν ανταποκρίνονται σε ακριβή στοιχεία. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι τα συστήματα του ελέγχου και της επιθεώρησης θα πρέπει να συμπληρωθούν και ενδεχομένως να αντικατασταθούν από συστήματα παρακολούθησης, ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ουσιαστικά βασίζονται σε κάποιες ε, πειραματικές και εμπειρικές ε, έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές και βασικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε και το κόστος της εγκατάστασης αυτών των συστημάτων. Μεταξύ 7 και 12.000 ευρώ είναι το κόστος, το ετήσιο κόστος για τα μεγάλα σκάφη και 1.500 με 2.500 για τα μικρότερα. Βεβαίως ε, μπορούμε να καλύψουμε τα πρόσωπα των ε, αλλιέων για να μην υπάρχει θέμα με τα προσωπικά δεδομένα. Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε ότι μπορεί κανείς να συγκρίνει τα στοιχεία που συλλέγονται από τις κάμερες, από στοιχεία τα οποία συλλέγουμε από άλλους αισθητήρε που επίσης βρίσκονται πάνω στα αλληλευτικά σκάφη. Συμπερασματικά θέλω να πω ότι ακριβώς ε, επειδή διαθέτουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες και όλες αυτές τις δυνατότητες παρακολούθησης εξ θα πρέπει να επιλέξουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνουμε σκάφη ε, διάφορων περιοχών και βεβαίως αυτό για να γίνει χρειάζεται προηγουμένως μία νομική εξουσιοδότηση, δημιουργία ενός πλαισίου νομικού έτσι ώστε να δοκιμάσουμε τα συστήματα αυτά, την τεχνολογία αυτή της εξαποστάσεως παρακολούθησης σε διάφορα σκάφη, διάφορες κατηγορίες σκαφών και διάφορες περιοχές. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η τροποποίηση του κανονισμού ελέγχου, του άρθρου 25 συγκεκριμένα α, προβλέπει την δυνατότητα εξοπλισμού των αληφτικών σκαφών με τέτοια συστήματα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ο βασικός κανονισμός, ο οποίος ισχύει σήμερα, προβλέπει ότι για να υπάρξει τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης χρειάζονται συγκεκριμένα ακριβά στοιχεία όσον αφορά όλες τις ε, εξόδους, όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα αλληλευτικά σκάφη έτσι ώστε να μπορούν να συγκρίνουμε τα στοιχεία και να έχουμε αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τους τρεις ε, πρώτους ε, ομιλητές ε, και μετά να δοθούν κάποιες απαντήσεις και συνέχεια να ακούσουμε και, άλλους, και άλλα μέλη. Οπότε η επόμενη ομιλήτρια είναι τώρα η Αντώνια Λιρόη. Από το Γραφείο Πολιτικής για την Ευρώπη του WWF. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να απευθυνθώ στην Επιτροπή Αλία σήμερα. Η παρουσίασή μου αφορά την παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω τις ε, προτεραιότητες που έχουν θέσει το VVF και κάποιες άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όμως θα συνεχίσω στα αγγλικά και θα κάνω την παρουσίαση στα αγγλικά. So first, why we need a revision? Because there is still remaining loopholes regularly reported, sometimes by χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό επειδή υπάρχουν πολλά παραθυράκια, αν θέλετε, στον νόμο, τα οποία ε, διαπιστώνουμε και εδώ βλέπετε για παράδειγμα ε, δύο περιπτώσεις οι οποίες έχουν ε, κοινοποιηθεί από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα παράνομες δραστηριότητε στην αγορά και εδώ αναφέρονται επίσης και οι αδυναμίες του συστήματος ελέγχου από το iWatch, το οποίο δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα σύστημα παρακολούθησης της λαθρείας παράνομης και άναρχης αλίας από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θέλουμε λοιπόν καλύτερους κανόνες ελέγχου έτσι ώστε να έχουμε ίσους κανόνες του παιχνιδιού ε, στο εσωτερικό των κρατών μελών για όλους τους αλληλείς. Θεωρούμε λοιπόν πως υπάρχουν δύο διαφορετικές διαστάσεις ε, του κανονισμού για τον έλεγχο της αλληλείας. Η μία διάσταση είναι η συγκέντρωση, διαχείριση και ανταλλαγή των δεδομένων σε, όλο το, σε όλη την αλυσίδα αν θέλετε, της ε, αλληλείας και για όλους τους αλληλείς, ενώ η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με την επιβολή της νομοθεσίας, δηλαδή ε, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά συστήματα ελέγχου και επιθεώρηση, ε, αποτρεπτικές κυρώσεις και διαφανείς πληροφορίε σε ό,τι αφορά την επιβολή της νομοθεσίας. Θα σας εξηγήσω λοιπόν το τι εμείς προτείνουμε σε ό,τι αφορά το νέο κανονισμό για τις απαιτήσει ελέγχων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν καταρχήν την πρώτη διάσταση, δηλαδή την συλλογή, τη διαχείριση και την ανταλλαγή των δεδομένων, θα πρέπει ε, να έχουμε, ε, να επιτύχουμε αλληλεία η οποία θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Τι σημαίνει αυτό, ότι καταρχήν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απομακρυσμένα συστήματα παρακολούθησης ε, και αυτό γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε την παρακολούθηση αλλά και επειδή οι κατανοητές θέλουν καλύτερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά ε, τα προϊόντα αλίας που καταναλώνουν. Άρα λοιπόν ε, υπάρχουν ε, συγκεκριμένα πλέον σε ό,τι αφορά τη χρήση απομακρυσμένων ε, συστημάτων παρακολούθησης σε όλα τα σκάφη. Για παράδειγμα, μία μελέτη από το 2017 του WWF με την χρήση βελτιωμένων τεχνολογιών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, σκάφη μεγαλύτερα από 15 ε, μέτρα ε, θα μπορούσε να είχε πολύ συγκεκριμένα πλειονοτήματα. Και βέβαια όλα αυτά τα συστήματα μπορεί να είναι προσαρμοσμένα σε κάθε διαφορετικό τύπο αλίας αλλά μπορούν να προσαρμοστούν σε όλους τους τύπους της αλίας και γι' αυτό θα χρειαστεί να έχουμε και σε ό,τι αφορά και την αλληλεία μικρή κλίμακα και την εραστεχνική αλληλεία, πλήρη συστήματα αναφορά των αλληλευμάτων. Άρα λοιπόν ε, υποστηρίζουμε την πρόταση τη Επιτροπή να υπάρξει εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και στη μικρή κλίμακα αλληλεία και στην ερασιτεχνική αλληλεία, με καταγραφή στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο όλων των λεπτομεριών σε ό,τι αφορά δηλαδή όλα τα αλληλεύματα, σε ό,τι αφορά τον τύπο, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και ούτω καθεξής. Ε, και επίσης ε, υποστηρίζουμε την ε, θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης και αδειοδότησης για όλους τους εραστέχνες αλληλείς και αντίστοιχη παρακολούθηση των δικών τους αλλιευμάτων στην, στις και στον Καναδά αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη και τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη παρακολούθηση με πιο θετική σχέση κόστους αποτελέσματος αυτό μπορεί ταυτόχρονα να ε, ε, βελτιώσει και, την, και την, ε, τις πιο, τα πιο πλήρη αλλά και αξιόπιστα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα. Ε, μπορούν με, αυτό, αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις, το περιβαλλοντικό αντίκτυπο και βελτιώνουν και την ανταπόκριση στις απαιτήσει της αγοράς σε ό,τι αφορά την καλύτερη διαφάνεια και την ε, λογοδοσία. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και για τους καταναλωτές να έχουμε καλύτερη ε, παρακολούθηση ό,τι αφορά τι αλευτικέ δραστηριότητε. Στο πλαίσιο λοιπόν τη αναθεώρησης του κανονισμού θα πρέπει ταυτόχρονα να βελτιώσουμε και την ιχνηλασιμότητα ε, των προϊόντων. Δηλαδή, για να σα δείξω εδώ στο χάρτη, τη σήμερα ημέρα εισάγουμε το 70% ε, των προϊόντων αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, παράγουμε μόνο το 30%. Αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε τις απαιτήσει σε ό,τι αφορά την εχνηρασιμότητα. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να ε, ε, βελτιώσουμε και τι απαιτήσει σε ό,τι αφορά τα σχετικά δεδομένα, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ε, πιστικό, πιστοποιητικό αλλιεύματο. Δηλαδή, να έχουμε μεγαλύτερο έυρος σε ό,τι αφορά τον αριθμό IMO. Θα πρέπει να έχουμε αναφορά και των μεθόδων αλλιέυσης και επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερο ορισμό των περιοχών αλίευσης ε, όπως για παράδειγμα ήδη εφαρμόζεται από την πλευρά άλλων χωρών όπω ε, οι ΗΠΑ. Τώρα περνάω στη διάσταση τη επιβολή τη νομοθεσία. Δηλαδή, καταρχήν γνωρίζουμε ότι μια νομοθεσία είναι τόσο αποτελεσματική όσο είναι η επιβολή τη. Οπότε, όπω ανέφερε και ο πλεγμένος ε, Επίτροπος Σενκεβίτσιους, η άλλη πλευρά του νομίσματος ε, του ελέγχου τη αλληλεία είναι η επιβολή της νομοθεσίας. Δηλαδή, ε, για να έχουμε βιώσιμη αλληλεία θα πρέπει να έχουμε να σεβαστούμε τη μεγάλη πλειοψηφία των αλλιέων οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, την, ε, μια καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να διευρύνουμε περισσότερο τον κατάλογο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα, ε, οι σοβαρές παραβιάσεις. Τι θέλουμε λοιπόν να περιληφθεί εδώ. Η απενεργοποίηση των αναμετατών του AIS, δηλαδή του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης. Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται σοβαρή παραβίαση το να μην πληρούνται οι υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την ε, μείωση των ε, περιπτώσεων αθέλητης ε, αλίευσης ευαίσθητων ειδών και επίσης οι περιπτώσεις όπου με κάποιο τρόπο συμμετέχουν οι αλληλείς παράνομη λαθρέα ή άναρχη αλληλεία, δηλαδή IUU. Επίσης, για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε περισσότερη και καλύτερη επιβολή τη νομοθεσία, θα χρειαστεί να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Δηλαδή, θα πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο του κανονισμού ε, εκθέσει ελέγχων, περιπτώσει παραβίαση, κυρώσει και ούτω καθεξής. Εμείς για παράδειγμα ζητήσαμε το 2017 και το 2018 πληροφορίες σε ό,τι αφορά αυτά τα στοιχεία και διαπιστώσαμε ότι είχαμε μόνο 1547 σοβαρέ παραβιάσεις που αναφέρθηκαν από τα κράτη-μέλη. Ε, και η συντριπτική πλειοψηφία όπως βλέπετε και στο γράφημα είναι στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και μόνο 449 από αυτέ τις 1547 περιπτώσει συνοδεύτηκαν από κυρώσει. Άρα λοιπόν τα μέτρα που έχουμε ε, επιβάλει μέχρι στιγμής είναι ε, δεν έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και δεν είναι δίκαιο το να αφορούν σε ένα ε, αριθμό λίγων μόνο κρατών μελών ε, περισσότερες από αυτές τις κυρώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, σοβαρή παρακολούθηση και επιβολή τη νομοθεσία με τι κατάλληλε κυρώσει, έτσι ώστε να έχουμε ίσους κανόνες του παιχνιδιού για τα ίδια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ολοκληρώνοντα λοιπόν εδώ να σας πω ε, το τι θα είναι σημαντικό για το WWF και για τις υπόλοιπες μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τους ελέγχους είναι το εξής. Θέλουμε να έχουμε πλήρως τεκμηριωμένη αλία με την ε, βοήθεια ε, των συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης. Θέλουμε όλα τα προϊόντα αλληλείας να είναι ειχνηλάσιμα με διαφανείς αλυσίδε αφοριασμού. Θα, θα πρέπει επίση να υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία σε ό,τι αφορά την επιβολή τη νομοθεσία, δηλαδή να έχουμε αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και αποτρεπτικέ κυρώσει και πρέπει να υπάρχει ένα ε, πλαίσιο ίδιων κανόνων, ίσων κανόνων του παιχνιδιού εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό αυτή, δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια σε το δικό μα position paper έχουν ε, συμμετάσχει μία σειρά από μη κυβερνητικέ οργανώσει που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ο κύριο Γιούγκερ Μπάτσλερ έχει ε, τον ε, λόγο από το Πανεπιστήμιο του Βάγκενίγκεν και συγκεκριμένα το τμήμα έρευνας του Βάγκενίγκεν. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στην έρευνα που κάνουμε στο πανεπιστήμιό μας, στο Wageningen. Είμαι ερευνητής και θα μιλήσω ιδιαίτερα για το σημείο 2, πώς δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάμερες και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα στα αλληλευτικά σκάφη για να βελτιώσουμε ε, και να εμβαθύνουμε την μέχρι τώρα έρευνά μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης χωρίς όμως να θεωρούμε ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο. Θα σας εξηγήσω καταρχήν πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα Έχουμε αλλιευτικά σκάφη τα οποία ε, ήδη είναι εξοπλισμένα με αισθητήρε και με κάμερες και μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα. Πρώτον, με εικόνες, με την συλλογή εικόνων οι οποίες στέλνονται σε ένα Ινστιτούτο, τις ε, παρακολουθούν, τις ε, αναλύουν και χρησιμοποιούν ε, ουσιαστικά το ημερολόγιο καταστρώματος σαν ε, συγκριτικό εργαλείο και μπορούν να συγκρίνουν τα στοιχεία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποιείται παντού στον κόσμο. Κοιτάξτε αυτό το χάρτη και παρακολουθείτε ότι υπάρχουν πειραματικές ε, χρήσεις αυτών των συστημάτων και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Υπάρχει ένας ε, μεγάλος αριθμός, 300-400 αλληλευτικά σκάφη, βλέπετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα σύγκρισης των στοιχείων και παρακολούθησης. Αυτό είναι για να δείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται για την συλλογή στοιχείων και για την βελτίωση της διαχείρισης ε, της ε, αλίας και των αποθεμάτων. Όσον αφορά τις εκφορτώσεις, μπορείτε να δείτε ότι έχουμε πολύ καλύτερες πληροφορίες, ε, πολύ πιο πλήρες και ακριβείς πληροφορίες. Όσον αφορά τις απορρίψεις, εκεί έχουμε ένα μεγάλο εράτηματικό σε πολλές από τις περιπτώσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς δηλαδή τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όσον αφορά τις απορρίψεις ε, στην ανοιχτή θάλασσα. Επιπλέον, αν κάποιος μπορεί να έχει κάμερες ε, που να συλλέγουν στοιχεία μπορούμε παραδείγματος χάρη να συγκρίνουμε κάποιες, κάποια δεδομένα όσον αφορά τις απορρίψεις και την επιβίωση των ε, αποθεμάτων. Μπορούμε δηλαδή να δούμε διαφορές μεταξύ των ε, αλλιευμάτων και των ε, εκφορτώσεων. Σήμερα τι κάνουμε. Στέλνουμε κάποιους επιθεωρητές στα αλλιευτικά σκάφη με ένα χαρτί και ένα μολύβι, οι οποίοι παρακολουθούν το τι συμβαίνει. σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πάρα πολύ ακριβή στοιχεία ή πρόκειται όμως για μία μέθοδο η οποία ουσιαστικά απαιτεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιθεωρητών. Τελικά βλέπουμε δηλαδή ότι μόνο το 5% των ε, αλλιευτικών σκαφών μπορούν να επιθεωρηθούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα πόσο αξιόπιστα είναι τα στοιχεία μας. Και γι' αυτό και ε, θεωρούμε ότι τα συστήματα παρακολούθησης ε, μέσω κάμερας είναι πολύ πιο ε, αξιόπιστα καθότι μπορεί να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό σκαφών. Μέσω κάμερας, μέσω συστημάτων GPS και βεβαίως παρακολουθώντας ε, την αλίευση αυτή καθεαυτή, τη διαλογή των αλιευμάτων και τις απορρίψεις. Κάποιος λοιπόν συλλέγοντας όλα αυτά τα στοιχεία, αυτές τις εικόνες μπορεί να τις αναλύσει, να τις συγκρίνει και να ελέγξει πώς ακριβώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Συνεχίζουμε παρόλα αυτά να στέλνουμε και επιθεωρητές επιτόπου στα αλλιευτικά σκάφη. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να συγκρίνει κατά πόσο η όλη διαδικασία και η παρακολούθηση μέσω της κάμερας είναι ακριβής. Στο παρόν ε, πειραματικό ερευνητικό πρόγραμμα έχουμε παρακολουθήσει τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις αλληλευτικών σκαφών, δοκότρατες και ήδη έχουμε προχωρήσει από το Μάιο του 2019 στην πράξη σε μια παρακολούθηση μέσω αυτών των συστημάτων. Κάποιος ο οποίος παραδείγματος χάρη έχει 100 διαφορετικά ταξίδια. Βλέπετε εδώ στη μαύρη γραμμή την παρακολούθηση. Δεν κάνουμε εδώ διαλογή βάση των ε, αποθεμάτων και των ειδών. Η παρακολούθηση γίνεται βάσει των εικόνων που μας ε, ε, στέλνουν. Αν θέλουμε όμως κάτι παραπάνω, περισσότερες πληροφορίες για ένα πολύ συγκεκριμένο είδος τόνου, σκουμπρί και παρακολουθούμε παραδείγματο χάρη τη μία ή την άλλη πλευρά του αλλιεύματος Πρόκειται για το κυλιδόβατο Σαλάχη. Και εδώ βλέπετε ότι η πιο στενή παρακολούθηση συγκρίνοντας αυτές τις εικόνες μας οδηγεί σε μια πολύ πιο ακριβή συλλογή στοιχείων. Βεβαίως αν αυτό γινόταν όπως καταλαβαίνετε σε όλα τα ε, ταξίδια των ελεκτικών σκαφών εδώ θα χρειαζόταν απεριόριστες ώρες υπάλληλοι οι οποίοι κάθονται στο γραφείο τους και συγκρίνουν συγκεκριμένες εικόνες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός και για στο πώς ε, συλλέγονται αυτές οι εικόνες. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ καθαρή η παρακολούθηση, οι κάμερες, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν τα είδη των αλλιευμάτων και να γίνονται οι μετρήσεις και οι συγκρίσεις με ακριβή και αξιόπιστο τρόπο. Επίσης, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το μέγεθος των αλλιευμάτων, γιατί αυτό βεβαίως ορίζει σημαντικά και τις απορρίψεις. Πρόκειται λοιπόν για μια πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα απαιτεί πάρα πολλές ώρες και εξαιρετικά πολλούς υπαλλήλους αν θέλουμε να καλύψουμε όλο τον ελληνικό στόλο. Και εδώ βλέπετε την εικόνα ενός σαλαχιού. Καταλαβαίνετε πόσες εικόνες περνάνε στο κομπιούτερ. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά αναγνωρίζουν τα είδη των ηχθείων και με αυτόν τον τρόπο Ξεκινήσαμε με ένα συγκεκριμένο ψάρι από τη μία και την άλλη πλευρά και φτάσαμε σε πιο περίπλοκες εικόνες πως ένα συγκεκριμένο ψάρι είναι στο, στη θάλασσα και πως ε, αλλάζει η εικόνα του όταν φτάσει πάνω στο σκάφος Και εδώ αναφερόμαστε στο είδος ε, αυτό το συγκεκριμένο τα πλατύψαρα. Η κάμερα ουσιαστικά λοιπόν καταφέρνει να εντοπίσει τα είδη των ε, ηχθείων με πάνω από 90% ακρίβεια. Έχουμε εδώ αυτά τα τρία είδη ψαριών τα οποία συγκρίνουμε και για τα οποία μπορεί ο υπολογιστής να ε, εντοπίσει με μεγάλη ακρίβεια. Εγώ πρέπει να σας πω που είμαι ειδικό για αυτό το είδος ψαριών. Δεν θα μπορούσα με αυτήν την ταχύτητα να κάνω ε, και να, φτάσω να κάνω ανάλυση των δεδομένων και να φτάσω σε αυτά τα αποτελέσματα. Όσον αφορά λοιπόν τα πλατήψαρα, έχουμε φτάσει μετά από έξι μήνες, από το Μάιο δηλαδή, σε εξαιρετικά ε, ακριβή αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τους αισθητήρε, τα δεδομένα που συλλέγουμε από τις κάμερες που βρίσκονται επί των αληθικών σκαφών κτλ. Αυτά έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τώρα με το ηλεκτρονικό αυτοσύστημα και την ανάλυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το θέμα τώρα είναι πώς οι πληροφορίες αυτές θα γίνονται όλο και πιο ακριβείς και πώς θα κάνουμε σε αυτά τα πειραματικά προγράμματα καλύτερη επιλογή δεδομένων για να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό βεβαίω, θα πρέπει να έχουμε την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξήσουμε υπερβολικά το φόρτο εργασίας και το ε, γραφειοκρατικό άχθος για όλους αυτούς που βρίσκονται στα αλληλευτικά σκάφη. Αυτό είναι μια προεπίθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου ή με τους συνεργάτες μου, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Έκανα λάθος με το όνομά σας, αλλά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλήρης παρουσίασή σας. Πάρα πολύ ωραία ήταν τα πρακτικά στοιχεία που δώσατε, αλλά εάν θέλαμε ε, να βάλουμε το ρέμι σε πάρα πολλά σκάφη, εκτός και αν έχει πραγματικά ανατρεπτικό στοιχείο και οδηγήσει σε πραγματική αύξηση ε, της ε, ε, αναφοράς του reporting μέσω των ηλεκτρονικών ε, στοιχείων καταγραφής και επιτήρησης ε, και οι καπετάνοι ας πούμε θα οδηγηθούν τελικά σε πιο ε, καλές σωστές πληροφορίες νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν έτσι διαζώσεις ας πούμε και διαγυμνού οφθαλμού να γίνουν αυτές οι επαληθεύσεις εάν θέλαμε να συμμορφωθούμε έγκαιρα με αυτό που προτείνει η Κομισιόν, θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Απάντηση. Είμαστε ακόμα στην αρχή και αν είμαστε τυχεροί θα μπορέσουμε τα επόμενα τρία χρόνια να συνεχίσουμε στην ανάπτυξη του συστήματος. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και μπορεί να εφαρμοστεί εάν υπάρχουν κάμερες ε, επιτόπου, πάνω στα σκάφη δηλαδή. Εάν όμως εξακολουθήσει να γίνεται ο έλεγχος χειρονακτικά και με συγκεκριμένες ε, λήψεις snapshots, και αν πρέπει χειρονακτικά ας πούμε να ελεγχθεί όλο το ταξίδι, πραγματικά δεν ξέρω πού θα βρείτε όλο τον κόσμο αυτό που θα πρέπει να κάθεται πίσω από έναν υπολογιστή όλη μέρα και να καταβάλει την προσπάθεια αυτή. Η δυνατότητα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε στο δικό μας Ινστιτούτο, γιατί εμείς το αναπτύξαμε αλλά έχουμε ας πούμε τέσσερα σκάφη. Αν θέλει κανείς να το εφαρμόσει σε δέκα σκάφη, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσλάβετε τους απαραίτητους που θα κάνουν αυτήν την ε, παρακολούθηση. Νομίζω ότι η διερεύνηση νέων ε, τεχνολογιών αυτή είναι η πιο αποτελεσματική λύση, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Πολύ ωραία. Ε, βέβαια ακούσαμε και στην πρώτη παρέμβαση του κυρίου Σαβουρέ ότι αυτά τα ε, μηχανήματα, ας πούμε αυτός ο εξοπλισμός όταν είναι πάνω στα πλοία μπορεί να δώσει πιο ασφαλή στοιχεία. Ακούσαμε λοιπόν τι είχε να μας πει ε, και ο κύριος Σαβουρέ και η κυρία Λερουά από την VVF. Φαίνεται ότι στην Ισπανία γίνονται πολλές παραβάσεις. Ε, δεν ξέρουμε όμως εάν πραγματικά παραβιάζουν μαζικά οι Ισπανοί ή εάν εφαρμόζουν καλά ε, και κατά γράμμα τους κανόνες, άρα οδηγούνται σε ε, μεγαλύτερο αριθμό διαπιστωμένων παραβάσεων. Το, το ζήτημα είναι να δούμε πραγματικά ποιο είναι το δυναμικό και πώς μπορούμε να επιτύχουμε το δυναμικό μας αυτό. Έχουμε ήδη πολλούς ε, εγγεγραμμένους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Μηγιαμών. Όχι, δεν ζήτησα το λόγο. Δεν ζήτησα το λόγο. Αλλά, παρόλα αυτά, ο κύριος Σαβουρέ μας είπε ότι έχουμε, θα έχουμε αυτές τις κάμερες ε, για τους ε, ε Έχουμε όμως χώρες όπως ε, η, Νέα Ζηλανδία που φαίνεται ότι έχει εφαρμόσει το σύστημα, η Νορβηγία, η Νέα Ζηλανδία ή άλλες έχουν επίσης και κάμερες σαν αυτές που προτείνει η Κομισιόν στο νέο κανονισμό ελέγχου ε, για να ε, ελέγχουν και την υποχρέωση αποβιβάς, ε, εκφορτώσεων. Αυτό θα μπορούσε να μας πει ο κύριος Σαβούρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί το Πανεπιστήμιο του Βάγκενιν μας έδωσε αυτήν την ε, αίσθηση ότι πρέπει να προσέξουμε και ε, βεβαίως ε, και οι ίδιοι θα πρέπει να δεχτούν τα συστήματα αυτά και να καταλάβουν πώς έχει η κατάσταση. Αλλά πέραν αυτού ρωτώ, ποια συστήματα ελέγχου ε, θα μπορούσαν να, χρησιμοποιούν, ε, και, να χρησιμοποιηθούν και επίσης ποιος θα πληρώσει το κόστος. Δεν κάτι το οποίο ε, κατά την άποψή μου δεν είναι πληρωτέο, δεν είναι και εφαρμόσιμο. Ωραία, άλλη μια ερώτηση. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε όλους όσοι μίλησαν σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με τους ε, στόχους της ΚΑΛΠ γιατί γι' αυτό ε, συζητάμε και γι' αυτό δουλεύουμε και πάνω σε αυτό με τον κανονισμό ελέγχου. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία μας περιέγραψε πάρα πολύ καλά τον κανονισμό ελέγχου. Όμως κάποια στιγμή στην παρέμβασή της ανα, είπε ότι θα πρέπει ε, να παρακολουθούμε το προϊόν μέχρι το μεταποιημένο προϊόν. Ε, πιστεύει η εκπρόσωπος Κομισιόν ότι μπορούμε να φτάσουμε όντως μέχρι τα μεταποιημένα, γιατί μέχρι τώρα δεν ε, καταφέραμε να προχωρήσουμε καθόλου όσον αφορά το θέμα αυτό και όσον αφορά τις ετικέτες και τη σήμανση προέλευσης. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και την ΕΦΚΑ για την τεράστια δουλειά που κάνει για τα συστήματα, τα συστήματα ελέγχου τώρα θα πρέπει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει βεβαίως να αναλυθεί και το κόστος και η αναλογικότητα ε, και αναρωτιέμαι μπορεί ο εκτελεστικός διευθυντής να μας δώσει την χρυσή γραμμή, πού βρίσκεται η χρυσή γραμμή ανάμεσα ε, στο κόστος και την ανάγκη επιτήρησης που θα φέρει αποτελέσματα. Τρίτον, στον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου να πω πρώτον ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εργασία που κάνουν. Ωστόσο, θεωρεί δυνατή, πιθανή την δυνατότητα μεγαλύτερης ε, εναρμόνισης ε, όχι μονάχα στα όσα προβλέπονται στο κανονισμό ελέγχου αλλά στα διάφορα συστήματα τα οποία έχουν προβλέψει οι μεμονωμένες χώρες για τον έλεγχο. Εναρμόνιση λοιπόν των ισχυών των συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου και αν κατά την άποψή του είναι αναλογικά σωστό το ε, να υπάρχουν παρατηρητές σε όλα τα σκάφη που θα κάνουν αυτόν τον έλεγχο όλου του αλλιεύματος και εάν εκείνοι ε, στην έρευνά τους έχουν παρατηρήσει ε, ποιου είδους μάλλον συνεργασία έχουν ε, είναι συνεργατικό σύστημα ή με κάποιο τρόπο μπορεί να δυσκολέψει την αλλιευτική δραστηριότητα των ιδίων των αλλιέων. Οπωσδήποτε, και αυτό είναι αμφισβήτητο, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε στρεβλώσεις καταστάσεις και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι για μια βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή αλία και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Έξι ερωτήματα ακούσαμε μέχρι τώρα. Ακούσαμε και τον κύριο Άσο και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο ε, στους ε, τρεις ε, πανελίσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ευχάριστο γεγονό ότι μπορούμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, θα ε, ήθελα να θέσω ερώτημα στον κύριο Μπασιλέρ. Τον ευχαριστούμε βέβαια για την παρουσίαση που έκανε σε σχέση με αυτό το σύστημα. Ε, και εγώ από αυτό που κατάλαβα ε, είναι ότι αυτό το σύστημα είναι κυρίω σύστημα διαχείριση ε, των αλευμάτων. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για του ίδιου ε, του αλληλεί. Δεν είναι ένα σύστημα δηλαδή κατεξοχήν ελέγχου, αλλά ε, κυρίω επιχειρησιακό, αν θέλετε, χαρακτήρα σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να θέσω εγώ τώρα σχετικά με αυτό είναι το εξή. Πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε τον, την προστασία τη ε, ιδιωτική σφαίρα, τη προσωπική σφαίρα των αλλαίων, γιατί είναι κάτι το σημαντικό για εκείνου. Δηλαδή, τι ακριβώ ε, θα γίνεται με αυτά τα δεδομένα, πού θα καταλήγουν, ε, πώς ε, θα διαχειριστούμε τα, ζητήματα, τα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτά τα δεδομένα. Ε, θα μπορούσε λοιπόν να μας πει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό ο κύριο Μπασιλέρ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εντάξει, δεν με πείθει πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα σε σχέση με την προστασία τη ιδιωτικότητα, ε, γιατί στις, ε, για παράδειγμα στα διάφορα εργοστάσια υπάρχουν κάμερε παντού. Τώρα στα ελευθερικά ποιο είναι το πρόβλημα. Εμεί εδώ που καθόμαστε δεν έχουμε κάμερε παντού. Λοιπόν, ε, κύριε Πατσέ, μπορείτε να ξεκινήσετε πάντω εσεί. Ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι το ότι συνεργαζόμαστε με τον κλάδο με τις επιχειρήσεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, τα δεδομένα δηλαδή τα οποία συλλέγουν οι κάμερες αυτές ε, βρίσκονται στην κυριότητα των ίδιων των αλλιέων. Δεν είμαστε εμείς δηλαδή που ε, είμαστε κύριοι αυτών των δεδομένων. Δεν, είναι στη δική μας ιδιοκτησία. Υπάρχει λοιπόν μία δήλωση ε, την οποία υπογράφουμε και με βάση την οποία οι αλλιείς μας επιτρέπουν να, χρησιμοποιήσουν, ε, να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα τους, δικά τους δεδομένα και μα επιτρέπουν να τα κάνουμε απλό, να τα φορτώσουμε δηλαδή στο δικό μα σύστημα. Τώρα το πώ αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο γενικότερα το νομοθετικό του ελέγχου τη αλίας δεν ξέρω ε, να σα πω γιατί βρίσκεται εκτό τη δική μου ε, σφαίρα, αν θέλετε ειδίκευση. Ε, πάντως εμείς συνεργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ πάντω ε, πω για να είναι ένα τέτοιο project ε, να στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά και βούληση από την των αλλαίων να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν. Δηλαδή, οι διάφοροι καπετάνοι έχουν τις, τα συστήματα καταστημένα στα σκάφη τους, έχουν τα δεδομένα αυτά και εμεί θα πρέπει να, να τρόπο να συνεργαστούμε μαζί τους. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη χρήση αυτών των δεδομένων για τους σκοπού του ελέγχου, δεν ξέρω να σα. πω. Υπάρχει ένα ερώτημα που δείχνει εκτός μικρόφωνου. Πάλι Δηλαδή μας λέτε ότι εάν οι ε, καπετάνοι ε, εάν δεν θέλουν να σας δώσουν τα δεδομένα ε, τότε δεν χρειάζεται να το κάνουν. Δηλαδή όλα αυτά τα, τα, τα χρήματα τα οποία δαπανώνται θα πηγαίνουν στον πρώτο. Αυτό μας λέτε. Ο κύριος Μπατσλέρ. Όχι. Υπογράφουμε μία δήλωση από κοινού με βάση την οποία μας παρέχουν αυτά τα δεδομένα. Οπότε Δηλαδή ε, υπογράφουν ότι ε, διατίθενται να συμμετάσχουν ε, στο συγκεκριμένο project και από εκεί και μετά είναι υποχρεωμένοι να μα τα διαβιβάζουν. Δεν ξέρω πώ θα γινόταν κάτι τέτοιο, πώ θα μεταφραστεί στο σύστημα ελέγχου. Ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα, κύριε Βατσέ, που έθεσε η κυρία άλλοι. Ναι, εμεί λοιπόν στο δικό μα το ίδρυμα δεν έχουμε ειδικού από τον τομέα του ελέγχου. Έχουμε επιστήμονε οι οποίοι εξετάζουν ακριβώ αυτά τα αλλιεύματα για να δούμε πώ μπορεί να γίνει η καταμέτρηση. Ε, και με του παρατηρητέ δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν ε, θετικότερε ε, περίοδο και αρνητικότερε. Δηλαδή, πριν από 20-30 χρόνια, οι δικοί μα ε, παρατηρητέ δεν ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι. Δεν, δεν είχαν δηλαδή θερμή υποδοχή στα αλληλευτικά σκάφη. Σήμερα μέρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και πράγματι ε, υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή. Ερώτημα του Προέδρου. Γιατί υπάρχει όμω καλύτερη αντιμετώπιση των παρατηρητών. Η απάντηση. Ναι, θεωρώ πω η συνεργασία ανάμεσα στον επιστημονικό, τον ελληνικό τομέα και τον κλάδο έχει βελτιωθεί. Δηλαδή, εγώ έχω ε, μιλήσει με πολλού καπετάνιου και γενικότερα προσώπου ε, του αλληλευτικού κλάδου ε, και έχουν διαπιστώσει πλέον και οι ίδιοι ότι ε, η επιστημονική πτυχή ε, μπορεί να βοηθήσει και του ίδιου. Δηλαδή, εμεί κάνουμε πολλά σε επίπεδο επιστημονική έρευνα και για παράδειγμα προσπαθούμε εδώ να επιτύχουμε περισσότερα σε ό,τι αφορά ε, την εκτίμηση του, του, των αποθεμάτων. Πράγμα το οποίο είναι θετικό. Δηλαδή, ε, μιλάμε για παράδειγμα για συγκεκριμένα αποθέματα για τα οποία ε, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα στη διάθεσή μας. Αν δούμε δηλαδή τα διαθέσιμα δεδομένα μας λένε ότι δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το απόθεμα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα σαλάκια αλλά οι ίδιοι αλληλεί μα λένε όχι, εμεί βλέπουμε τεράστιε ποσότητε SLH. Οπότε ακριβώ σε αυτό έγκυται η χρησιμότητα τη συνεργασία, ότι μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα. Ο ε, ε, επιστημονικό τομέα με τον αλληλευτικό τομέα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ πω ε, πλέον είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη στα σκάφη οι επιστήμονε. κύριε Σαμπουρέ, λέει ο πρόεδρο, οι δικοί σα επιθεωρητέ συμφωνούν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, έχει βελτιωθεί η συνεργασία. I Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε διάφορες περιπτώσεις αρνητικής αντίδρασης, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου συνεργάζεται μαζί μας. Όσον αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης, θέλω να απαντήσω στην κυρία Μπιλμπάου Βαρντικά που έκανε μια ερώτηση επ' αυτού. Κοιτάξτε, όντως και εμείς βασιζόμαστε στην αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει καταρχήν να κοιτάξουμε τα δύο πιο υψηλά επίπεδα ε, κινδύνου όσον αφορά τις κατηγορίες των ε, αλλιέων και των αλλιευμάτων. Δηλαδή να εξοπλίσουμε στην πρώτη φάση, σε αυτή την πειραματική φάση, κυρίως τα αλλιευτικά σκάφη που έχουν χαρακτηριστεί σαν υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου σε αυτές τις κατηγορίες καφών και να παρακολουθήσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν προετοιμαστεί από κοινού με την Επιτροπή μετά από πολλή ε, προετοιμασία και ανάλυση αυτών των συστημάτων εξ παρακολούθησης της αλίας. Σε αυτές τις κατευθυντηρίες γραμμές, σε αυτές τις οδηγίες, έχουμε ήδη κάνει μια ανάλυση και για το κόστος ε, και για τις διάφορες κατηγορίες αλληλευτικών σκαφών. Όπως σας είπα, το κόστος είναι μεταξύ 7 και 12.000 ευρώ ετήσιο κόστος ανάλογα με το Σκάφος, το μέγεθος του σκάφους και το λειτουργικό κόστος ε, περίπου 2 με 2.500 ευρώ το χρόνο. Πιστεύω ότι αυτό το κόστος μπορεί να καλυφθεί, βεβαίως αυτό εξαρτάται και από την απόφαση των κρατών μελών και αυτό θα ληφθεί σε εθνικό επίπεδο ε, από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά βεβαίως πρόκειται για απόφαση που εξαρτάται και από τα κράτη. Τώρα, η προστασία της ε, ιδιωτικότητας. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα προστασίας της ιδιωτικότητας. Το θέμα είναι για ποιο χώρο συγκεκριμένα θέλουμε να υπάρξει αυτή η προστασία. Επαγγελματικό χώρος, προσωπικά δεδομένα και συμφωνώ με τον συνάδελφο από την Ολλανδία ότι θα πρέπει το σύστημα να λειτουργεί σωστά, να υπάρχει σωστή συντήρηση και αυτό βεβαίως είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση του καπετάνιου, του πλειοκτήτη, αλλά και βεβαίως τον, του πληρώματος. Γιατί από αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ακρίβεια των στοιχείων. πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση ε, για αυτά τα συστήματα εξ αποστάσεως τηλεπικοινωνίας, όπως έχουμε και με άλλα συστήματα EMS, συστήματα συλλογής πληροφοριών σε άλλα συστήματα με τα οποία έχουμε εξοπλίσει τα σκάφη. Θα ήθελα εδώ να πω επίσης και να υπογραμμίσω ότι περνάμε από μία αλλιευτική πολιτική και τον έλεγχό της σε μία που βασίζεται στον έλεγχο και στην παρακολούθηση, σε μία αλλιευτική πολιτική που βασίζεται στην ε, παρακολούθηση μέσω αυτών των συστημάτων και γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει μία ευαισθητοποίηση του κλάδου, να πείσουμε δηλαδή όλους αυτούς που συμμετέχουν ότι αυτό το νέο σύστημα είναι καλύτερο για αυτούς. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις πριν επανέλθουμε στους ομιλητές. Κυρία Σάλιβαν, έχω για τον κύριο Σαμπουρέ μια ερώτηση. Ποιες είναι οι αποκλήσεις, οι εξαιρέσεις όσον αφορά τα δεδομένα που σήμερα υπάρχουν, τις οποίες θέλετε να υπάρξει τροποποίηση για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, καλύτερη παρακολούθηση. Τι τροποποίησεις δηλαδή προτείνετε εσείς για να αλλάξει η κατάσταση και να είναι πιο αποτελεσματική παρακολούθηση. για την Ισπανία, για τις παραβιάσεις, αυτό δηλαδή που αναφερθήκατε, υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές στα στοιχεία ε, μεταξύ του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Πώς μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση στις κυρώσεις και στην ε, εφαρμογή γενικότερα, ιδιαίτερα για τις χώρες αυτές όπου παρακολουθούνται παρακολουθούμε ακόμα να υπάρχουν συγκεκριμένες παραβιάσεις, μεγάλος αριθμός παραβιάσεων. Επίσης έχω μία ερώτηση για το μέγεθος των σκαφών στα οποία έχετε εγκαταστήσει τέτοιες κάμερες. Μιλάμε συνεχώς για βιώσιμη αλληλεία, ότι θέλουμε να στηρίξουμε την τοπική κοινότητα και την τοπική αλληλευτική δραστηριότητα. Ρωτάω λοιπόν, αυτή η τεχνολογία την οποία προτείνεται μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει και σε πολύ μικρά σκάφη. Ε, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση απευθύνεται στον Ολλανδό συνάδελφο. κυρία Λερόη ο κύριο Σαβουρέ για την Ιταλία, την Ισπανία και τις χώρες με μεγάλες παραβιάσεις και κυρώσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή η ακρόαση που αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης θα λάβει χώρα στις 2 Δεκεμβρίου. Μα εδώ πρόκειται για ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα και γιατί επιλέξαμε αυτές τις ημερομηνίες και αυτή τη σειρά για τις ακροάσεις. Πραγματικά, αν αυτό το επιβάλλουμε και στα μικρά αλλιευτικά σκάφη, Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το θέμα των λεγόμενων choke spaces, των ειδών αυτών και το θέμα της ε, υπεραλίευσης. νομίζω ότι αυτό έχει εκλείψει από τη Βόρεια Θάλασσα. Έχουμε καλύψει όλες ε, τις, όλα τα είδη, ακόμα και τον γάδο και νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι το παράδειγμα της Βόρειας Θάλασσας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Κύριε Πρόεδρε, έχω και μία ερώτηση που θέλω να απευθύνω στην ε, Επιτροπή. Γιατί δεν ε, σταματάτε τη διαδικασία εδώ. Ακούσαμε αυτόν τον εξαιρετικό εμπειρογνώμονα από το Πανεπιστήμιο, ερευνητή από το Πανεπιστήμιο του Βάγκενιγκεν, ο οποίος σας δίνει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την εγκατάσταση κάμερας στα αλλιευτικά σκάφη. Γιατί λοιπόν να μην αναπτύξουμε μια τέτοια τεχνολογία η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανάγκες μπορούμε ενδεχομένως να βρούμε άλλου είδους και πολύ πιο αποτελεσματικές ε, λύσεις. Κυρία Αμάτο, αναλογικότητα και ασφάλεια ποινή. Ε, ε, αν δεν καθορίσουμε τα δύο στοιχεία αυτά, τίποτα δεν θα καταφέρουμε με τούτο τον κανονισμό που αφορά τους ελέγχους. Επίσης, δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει από τους εμπειρογνώμονες, ρωτώ, αν πρέπει να ξεχωριστούν τα διάφορα τμήματα του στόλου. Νομίζω ότι δεν θέλουμε, ε, και όλοι συμφωνούμε σε αυτό, να μην συνθλίψουμε τους ε, αλείς από την γραφειοκρατία. Ε, είτε είναι μικρά, είτε είναι μεγάλα σκάφη, είτε είναι κάτω από 12 μέτρα όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει κάποια φορά σε μια διαδικασία, ακόμα και ο ίδιος που έχουν τρία-πέντε ε, άτομα πλήρωμα, ε, ακόμα και ο καπετάνιος, ο σκίπερ, αν και στα Ιταλικά όταν λέμε σκίπερ εννοούμε πιο πολύ τα γιότ και τα σκάφη αναψυχής. Εν πάση περιπτώσει, οι καπετάνιοι κάνουν τα πάντα. Εγώ σας καλώ πραγματικά να ε, βρεθείτε με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και ταπεινότητα σε ένα σκάφος, να καταλάβετε ξέρετε τι γίνεται. Πάτε λίγο σε ένα αλλιευτικό σκάφος, μείνετε 14 ώρες, καμιά φορά και περισσότερες ώρες ε, μεσοπέλαγα για να δείτε τι συμβαίνει γιατί διαφορετικά μιλάμε για καθαρή θεωρία. Βεβαίως είναι καλοδεχούμενοι οι ερευνητές. Εγώ δεν βλέπω τόσο μεγάλη, δεν διαπιστώνω τόσο μεγάλη εχθρότητα από τους αλληλεί. γιατί ε, μιλάμε συνέχεια για καθαρή δουλειά, για γαλάζια οικονομία κτλ. Μιλάμε για διαρκή επιτήρηση, ε, αλλά δεν είμαστε καν ε, σε θέση να επιτηρήσουμε και να ελέγξουμε τις μεγάλες μολυντικές βιομηχανίες και τελικά ε, πέφτουμε πάνω στους απλούς μικρούς αλείς. Όσον αφορά την Ιταλία και την Ισπανία, ακούγεται ότι έχουν περισσότερε περισσότερες παραβάσεις. Εγώ έκανα την ερώτηση γιατί έχουμε περισσότερους ε, ας πούμε παραβάτες. Μα γιατί ε, γίνεται κοινοποίηση των ελέγχων. Ε, όσον αφορά τους ελέγχους, ε, θα ήθελα να, σας, ε, να δείτε πώς αυτό το σύστημα των points δεν εξυγχρονίζεται με τον ίδιο τρόπο και εξωτερικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πολλές χώρες σημαντικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι πρόκειται για κανονισμό, δεν τον υλοποιούν, δεν τον εφαρμόζουν. Είναι κανονισμός, δεν, πρέπει απλώς να εφαρμοστεί, δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Όσον αφορά την κυρία του VVF, ε, ε, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει εδώ τόσο πολύ η ίχνη λασιμότητα. Θέλω να πω, ε, κυρίως τα μεγάλα μαγαζιά ξέρουμε ότι ξέρουμε ε, ότι πολλές φορές ε, τα λεύματα που προσφέρουν ε, έχουν, έχουν αλλιευθεί ας πούμε εκτός των συνόρων. Ξέρουμε αν έχει υπάρξει κοινωνικό dumping, ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι. Uh, ναι. Ε, αντιλαμβάνομαι αυτά που είπε η συνάδελφος μόλις τώρα και πραγματικά και εγώ βρισκόμαστε σε σύγχυση. Δηλαδή, ακούμε ότι ε, ε, υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα, δηλαδή σε ό,τι αφορά Ιταλία και Ισπανία βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσει παραβιάσεων, ενώ σε άλλες όχι. Και χθε είδαμε ένα γράφημα όπου μας ε, έδειξε ότι οι περισσότερες από τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους λαμβάνουν χώρα στη Βόρεια Θόλασσα. Οπότε πραγματικά χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα και χρειαζόμαστε πιο αξιόπιστα από όλα τα κράτη-μέλη, από όλες τις περιοχές, για όλες τις παραβάσεις, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχει σε διαφορετική περίπτωση νόημα να προχωρήσουμε περισσότερο. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Και η ε, ε, Υπηρεσία ε, Ελέγχου της και η Επιτροπή και όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης, Είναι προβληματικό επίση το ότι όπω όπως είδαμε δηλαδή, κάποια κράτη-μέλη για τα οποία βλέπουμε πολλέ παραβιάσει, ενώ για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν βλέπουμε τίποτα. Οπότε δεν ξέρουμε εκεί τι συμβαίνει σε επίπεδο παραβιάσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, θέλουμε να ε, ξεφύγουμε από ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στη δειγματοληψία και θέλουμε να κινηθούμε προ ένα σύστημα με πιο συστηματική παρακολούθηση, ε, τότε ε, θα συμφωνήσω με αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι ενδεχομένω να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην πράξη ένα τέτοιο συστηματικό ε, σύστημα παρακολούθηση, δηλαδή μόνιμης παρακολούθηση, ή δεν θα αξίζει από πλευρά σε κόστου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε ε, ε, να, να έρθουμε σε επαφή με τα χώρε εκείνες που ήδη έχουν εφαρμόσει αυτό το σύστημα για να δούμε ποιο είναι το, το όφελος, ποιο είναι το κόστος, ποιος αναλαμβάνει το να καταβάλει αυτές τις δαπάνες και τι συμβαίνει ακριβώς με τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παραβιάσεις. Δηλαδή η καλύτερη τεχνολογία δεν σημαίνει αυτόματος θα υπάρχουν λιγότερες παραβιάσεις γιατί υπάρχουν μία σειρά από διαφορετικοί τρόποι ε, του να κοροϊδέψει αν θέλετε κανείς ε, τη νέα τεχνολογία και να συνεχίσει να προβαίνει σε παραβιάσεις. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε άλλα μέρη του κόσμου, τότε ε, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος από αυτές τις χώρες που ήδη το εφαρμόζουν για να μας πει πώς εφαρμόζεται, ποιο είναι το όφελος, ε, ποια είναι τα προβλήματα. Θα ήταν δηλαδή πάρα πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Φεραντίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Φεραντίνο, όσον αφορά την ιδιωτικότητα ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Να σας πω ότι και στην Ιταλία ε, ο κλάδος και μέσω των οργανώσεων εκφράζει πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις όσον αφορά ε, τις κάμερες κλειστού κυκλώματος. Εγώ δεν λέω ότι ε, ε, εάν αυτές οι κάμερες αφορούν μονάχα ένα συγκεκριμένο κομμάτι του σκάφους ότι δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά την ιδιωτικότητα. Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν πριν εφαρμόσει ε, υποχρεώσεις προς τους ε, αλληλείς ε, και πριν τους οδηγήσει σε επιπλέον κόστος, τότε θα πρέπει η Κομισιόν, την καλό λέω, να προσέξει και να, να μιλήσει περισσότερο με τους αλληλείς, γιατί οι περισσότεροι ψαράδες κερδίζουν τα χρήματά τους και τη ζωή τους με πάρα πολύ σωστό και νόμιμο τρόπο. Στις τρίτες χώρες που ε, διαπιστώνονται οι μεγαλύτερες απάτες καθώς επίσης ε, και ε, οι μεγαλύτερες παραβιάσεις ε, περιβαλλοντικές, εργασιακές κλπ. Εκεί καθορίζουμε, βλέπουμε ότι έχουμε τόσο αυτούς τους κανόνες που δεν εφαρμόζονται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής επίσης ή βεβαίως να έχουμε κανόνες που να τους επιβάλλουμε τους κανόνες στους αλληλείς της Ευρώπης αλλά να μην στραβλώνουμε τον ανταγωνισμό η χνηλασιμότητα είναι πολύ σημαντικό για τα, τα ήδη. Ε, θα πρέπει ε, στις συσκευασίες ε, να αναφέρονται όλες, όλα τα αλλιεύματα καθώς επίσης και όλες οι παρτίδες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψουμε τους καταναλωτές. Μπορούν να υπάρξουν λύσεις οι οποίες ενδεχομένως να εγείρουν ε, την, ε, ε, οι οποίες να καθησυχάζουν τους καταναλωτές χωρίς όμως να σημαίνουν και υπερβολικό φόρτο για, την, για τον κλάδο. Ευχαριστώ η κυρία Αγγιλέρα. Καλημέρα σε όλους. Εγώ είμαι η συγγήτρια για αυτόν τον κανονισμό ελέγχου και θα ήθελα ε, να μιλήσω στο τέλος, αλλά μια και ξεκίνησε νωρίς η συζήτηση, θα κάνω κι εγώ κάποιες, κάποια σχόλια, θα υποβάλω κάποιες ερωτήσεις που προέκυψαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, το, αυτό το πιλωτικό ε, του Πανεπιστημίου, αλλά είναι πιλωτικό. Το λέω, το τονίζω. Εμείς το ζητήσαμε, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που χρειάζεται τουλάχιστον τρία επιπλέον χρόνια. Και οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα αυτό για να δούμε αν μπορούμε ε, να πάρουμε κάποια στοιχεία του συγκεκριμένα. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι αμφισβήτητο. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει ε, ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εμείς στα χέρια μας έχουμε όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ε, ε, μια συγκεκριμένη πρόταση, ένα συγκεκριμένο κανονισμό δεν προχώρησε, δεν ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη θητεία, θα προχωρήσει σε τούτη εδώ. Θα παρουσιαστεί η έκθεση το Φεβρουάριο και ήδη ξαναρχίζουμε όλες τις συζητήσεις, μετροπολογίες κλπ και δεν ξέρω εάν πραγματικά θα έχουμε το χρόνο για να αξιολογήσουμε σωστά τέτοια πιλωτικά τόσο ενδιαφέροντα προγράμματα πολλές ερωτήσεις και γενικώ έτσι ασάφεια σχετικά με τα αποτελέσματα ε, στην Ισπανία και την Ιταλία. Μας αυτές τις χώρες γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και ε, επιβάλλονται περισσότερες κυρώσεις. Άλλοι ελέγχουν λιγότερο, επιβάλλουν κυρώσεις λιγότερο. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε. Καμιά φορά είστε ηρωνικός. Ε, βέβαια είναι ευγενής η ηρωνία σας όταν λέτε τι γίνεται στην Ισπανία. Θα σας πω εγώ τι γίνεται στην Ισπανία. Ελέγχονται καλύτερα περισσότερο τα πράγματα. Αυτό είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Αυτό που πρέπει είναι να έχουμε καλύτερο κανονισμό, καλύτερη, μεγαλύτερη εναρμόνιση έτσι ώστε ε, να μην υπάρχει περιθώριο διακριτικής μεταχείρισης και επίσης να μην επαφίεται ε, είτε στο πολιτικό κριτήριο μιας κυβέρνησης είτε στον υπερβάλλοντα ζήλο ενός ε, δημοσίου υπαλλήλου. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε αυτή την εναρμόνιση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, προς Θεού και εγώ τώρα άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό και καταλαβαίνω ότι καθόλου εύκολο δεν είναι. Ωστόσο αυτή η ε, απλούστευση, αυτή η θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και τα θέματα και να λάβουμε υπόψη μας και την μικρή κλίμακα αλληλεία και την ερασιτεχνική. Είτε θα τα κάνουμε τα πράγματα σοβαρά, είτε δεν μην τα κάνουμε καθόλου. Πρέπει οπωσδήποτε η εναρμόνιση να προχωρήσει και θα πρέπει να επιτύχουμε κάτι το οποίο θα είναι εφικτό αλλά για όλους. Θα είναι εφικτό, δυνατό για όλους. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πασκάλ Σαβουρέ, ε, γιατί νομίζω ότι η υπηρεσία αυτή έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να τον παίξει αυτό το σημαντικό ρόλο. Πιστεύω όμως ότι η ΕΦΚΑ, εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα απαιτούνται σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτήν την εναρμόνωση. εναρμόνωση. Εάν εντωμεταξύ καταφέρουμε να έχουμε μια, ε, ένα καλό κείμενο εναρμονισμένο για όλους θα πρέπει και η ΕΦΚΑ οπωσδήποτε να διευρύνει το ρόλο της έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό περισσότερα, περισσότερους πόρους, οικονομικούς και άλλους, περισσότερα μέσα, γιατί διαφορετικά η ΕΦΚΑ δεν θα μπορέσει αποτελεσματικά να κάνει την ε, δουλειά που πρέπει να κάνει. Επομένως, ρωτώ τον Διευθυντή με ένα νέο εναρμονισμένο για όλους κανονισμό, η ΕΦΚΑ θα μπορούσε να καλύψει έτσι όπως έχει σήμερα ε, τις νέες απαιτήσεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει λίγο η δομή της. Τελειώνω με το εξής. Όλα αυτά που ακούσαμε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα μας βοηθήσουν και οπωσδήποτε ξεκαθαρίστηκαν πολλά θέματα. Το πρόβλημα που έχουμε με την ψηφιοποίηση είναι η μετέπειτα εξελίξεις, ε, γιατί σε snapshot δεν μπορούμε να δούμε την εξέλιξη. 30 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, μόνο ο Αντιπρόεδρος. Ναι, νομίζω πως είναι σωστό αυτό που υπόθηκε, ότι δεν θέλουμε ε, να λαμβάνει χώρα απάτη. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το σημερινό σύστημα δεν λειτουργεί σήμερα. Οπότε με, ε, με τρομοκρατεί λίγο αυτή η ιδέα της Επιτροπής ότι κάθε ψάρι που θα βγαίνει από τη θάλασσα θα πρέπει να καταμετράται γιατί ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν πάρα πολύ ακριβό. Και ποιο ακριβώς θα καταβάλει το ε, κόστος για αυτό το ιδιαίτερα ακριβό σύστημα. Δηλαδή σίγουρα μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις, αλλά εάν ακολουθήσουμε αυτή την ιδέα της Επιτροπής ότι θα πρέπει να καταμετράτε κάθε ψάρι που αλλιεύεται, πραγματικά κάτι τέτοιο θα ήταν λανθασμένο και θα επιβαρύνει πάρα πολύ και τους αντιήσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ε, απευθύνομαι στους ε, ομιλητέ λοιπόν του πρώτου πάνελ. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που αναφέρθηκαν. Κύριε Σαβουρέ, εσείς αναφέρθηκατε σε μια σειρά από διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Και ειδικότερα εδώ βέβαια εστιάζουμε κυρίως στις ε, κάμερες. Επίσης αναφέρθηκε και το ζήτημα του μεγέθους των σκαφών. Εσείς είπατε ότι ε, θα ξεκινήσουμε από τα μεγαλύτερα σκάφη και εκείνα που είναι τα πιο έποπτα, αν θέλετε, για περίπτωση παραβίαση, σε εκείνα όπου θα μπορούσαν να σημειωθούν τα περισσότερα προβλήματα. Και επίση αναφέρεται και το ζήτημα των περισσότερων παραβιάσεων που παρατηρήθηκαν στην Ισπανία και την Ιταλία μόνο και όχι σε άλλα κράτη-μέλη. Μήπω μπορείτε να δώσετε απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο ε, Σαβουρέ. Ίσως ε, δεν ήμουν ξεκάθαρο σε αυτά που είπα, αλλά δεν είπα ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος του σκάφους αφενός ε, και το μέγεθος του κινδύνου αφετέρου. Έχουμε μια αξιολόγηση του κινδύνου σε ό,τι αφορά ε, το, ε, το μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά και τον αντίκτυπο ε, και σε γενικέ γραμμέ τα μεγαλύτερα σκάφη μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο αλλά μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει και ένα μικρό σκάφο. Εμεί εδώ είπαμε ότι εξετάζουμε, κάνουμε δηλαδή τη συνέρευνά μα ανα segments, ανα συγκεκριμένου τομεί. Εξετάζουμε για παράδειγμα πέραν του μεγέθου του σκάφου και το είδο των εργαλείων, την εποχικότητα τη αλίευση, το είδο του, του, του αλλιεύματο και ούτω καθεσής. Άρα λοιπόν ένα σύστημα RM θα μπορούσε να ε, προσαρμοστεί και για κατάσταση σε ε, πολύ μικρά σκάφη όταν δηλαδή θα έχουμε φτάσει ε, στα πιο εξελιγμένα επίπεδα της στρατηγικής διαχείρισης κίνδυνων μας. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα σε ό,τι αφορά ε, αυτές τις ε, αλευτικέ δραστηριότητε ε, θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο ποιο είναι το πλαίσιο αυτού του project. Υπήρχαμε δηλαδή δύο project, το ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα στη Σκωτία, το οποίο είχε την, ένα σύστημα επιστώσεων για αλλιεύματα δηλαδή παροχή υψηλότερων ποσοστώσεων για του αλληλεί εκείνου ε, που ε, δήλωσαν διατεθειμένοι να αποδεχτούν την εγκατάσταση ενό συστήματο άδεια στο σκάφο του. Ε, και αυτό το πρώτο πιλωτικό project οδήγησε μια κατάσταση που παρότι δεν υπήρχε ένα πλαίσιο επιβολής της νομοθεσίας, παρόλα αυτά οδήγησε σε κάποια δεδομένα. Και από εκεί και μετά υπήρξε και το πρόσωπο από την πλευρά της ε, ε Ισπανικής Υπηρεσίας ε, Ελέγχου της Αλίας. Η, ε, η Αγγλία επίσης προέβησε ένα τέτοιο πιλωτικό σύστημα, ενώ από τις χώρες της υπηρετικής Ευρώπης η Δανία διεξήγαγε ένα τέτοιο πιλωτικό project για κάποια χρόνια με 11-12 αν με αλληλευτικά σκάφη. Ε, αυτές λοιπόν οι βέλτιστε ε, πρακτικές θα μπορούσαν να μελετηθούν ε, περαιτέρα και με βάση αυτέ θα μπορούσαμε να προτείνουμε ένα πρώτο σετ, μια πρώτη δέσμη κατευθυντηριών γραμμών. Βρισκόμαστε ακόμα βέβαια στι πρώτε φάσει ακριβώ του πειραματισμού με τέτοιου είδου ε, συστήματα και όπω το ανέφερε και ο συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο του Βάγκενιγκεν, ακολουθούμε ακόμα περισσότερο την προσέγγιση με βάση τον έλεγχο και την επιθεώρηση, όχι την καταμέτρηση. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα ε, την ε, αναθεώρηση του κανονισμού σε σχέση με τον έλεγχο και τον ρόλο της ΕΦΚΑ, νομίζω πως αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι εμείς θα έχουμε αναλάβει σε εκείνο το πλαίσιο τον ρόλο ενός επιθεωρητή σε ό,τι αφορά τα ενωσιακά ύδατα. Αυτή τη στιγμή δεν το κάνω, το κάνω σε ε, ύδατα τρίτων χώρων. Πάντως, ε, αυτό που θα συζητηθεί μέσα στους επόμενους ε, μήνες είναι η επιλεξιμότητα των κοντιλίων για τους ελέγχους που θα περιληφθούν μέσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Ελίας και στα υπόλοιπα ταμεία για την Αλία. Ε, αυτή λοιπόν η ένταξη των σχετικών επόρων μέσα στο, στα σχετικά ταμεία θα είναι μια πολύ, ε, μια πολύ σημαντική συμπληρωματική υποστήριξη. Μια υποστήριξη βέβαια η οποία δεν θα απορροφηθεί από την ίδια την ΕΦΚΑ αλλά ουσιαστικά θα μεταφερθεί στα ίδια τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των ελέγχων τους. Κάτι ακόμα που θα ήταν σημαντικό για το σύστημα επιθεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπάρξει ένα κοινό σύστημα πιστοποίησης ε, ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει ένα, να υπάρχουν ίσοι κανόνε του παιχνιδιού, αν θέλετε, για όλο τον κλάδο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι και επιθεωρήσει. σε ό,τι αφορά ε, τις παραβιάσεις που παρατηρούνται στη Μεσόγειο και ειδικότερα στα κράτη-μέλη Ισπανία και Ιταλία, όπως ήδη είπα, είναι, ε, ε, έχουμε ένα όραμα το οποίο βασίζεται στην εφαρμογή από όλους και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να ε, ε συλλέγουμε στοιχεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ε, για, σε, για είδη τα οποία έχουν ε, περιληφθεί ε, στον κανονισμό GDP και ειδικότερα δηλαδή σε με, είδη όπως ο ερυθρός τόνος και κάποια άλλα είδη τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στη σύσταση του GFCM. Άρα δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πλήρη δεδομένα, μια συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά όλα τα είδη τα οποία αλλιεύονται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επιλεκτικά δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα για τι παραβιάσει. Ελπίζω να κάλυψα όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Σίγουρα από τη ε, δική μα ε, πλευρά τη Επιτροπή, δηλαδή, θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη τη ΕΦΚΑ στη φάση δηλαδή τη υποβολή ανθρωπολογιών που θα υποβάλουμε εμεί σε σχέση με την πρόταση που θα κάνει η Επιτροπή για την αναθεώρηση του κανονισμού. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα γαλλικά. Όσον αφορά την Ιταλία και την Ισπανία, υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι. Το ερώτημα είναι αν αυτό αντιστοιχεί και στον αριθμό των αλλιευτικών σκαφών. Αυτό που μπορώ να απαντήσω καταρχήν είναι ότι όσον αφορά την πιστοποίηση ISO 1000 15 η πιστοποίηση στην Ισπανία έχει προοδεύσει πάρα πολύ σημαντικά και μάλιστα από μέρους της α, ίδιας της χώρας, των εθνικών αρχών, του Υπουργείου, παραδείγματος χάρη, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό και ζητάμε μεγάλη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Είδαμε επίσης και στην εφαρμογή του συστήματος των κυρώσεων για τις πολύ σοβαρές παραβιάσεις ότι υπάρχει υποχρέωση να γίνει και μια νομοθετική μεταρρύθμιση. Ας πούμε στην Ιρλανδία υπάρχει θέμα, πρέπει να υπάρξει συνταγματική μεταρρύθμιση. Όλα αυτά λοιπόν κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια. Υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης της ε, πληροφορίας και στα δεδομένα. Πολλές φορές ε, προσκρούμε είτε σε προβλήματα πολιτικής βούλησης, είτε σε άλλου είδους ε, εμπόδια. Και όλα αυτά, εξαρτάται από τη χώρα βέβαια, θα πρέπει να ξεπεραστούν. Το θέμα τώρα του κοινωνικού ντάμπινγκ και της χνασιμότητας, το πώς μπορούμε δηλαδή να βρούμε τις πραγματικές αιτίες. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά αλλιευμάτων, τα catching certificates, τα επίπεδα. Όσον αφορά τον εκτελεστικό κανονισμό, ξέρουμε ότι παγκοσμίως, όσον αφορά τον αριθμό του IMO, του Παγκόσμιο Οργανισμό της Θάλασσας, ο κανόνας είναι 15 μέτρα. Και από τη στιγμή που θα τηρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον κανονισμό αυτό και το ψήφισμα του 2017 για τον αριθμό του IMO, και όταν συμπεριλάβουμε και όλες τις σημαίες ευκαιρίας και όλα αυτά που πρέπει να συμπεριλάβουμε για να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό dumping και ευθυγραμμιστούμε με τους διεθνείς κανόνες, θα μπορούμε να έχουμε πιο πολύ διαφάνεια. Υπάρχουν εδώ και οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, κάτι βεβαίως που θα μας οδηγήσει σε άλλες ε, συζητήσεις για πιο συνεκτική πολιτική σε κοινωνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Ναι. Όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Σάλιβαν. Ναι, εμείς έχουμε τρία σκάφη, 40 μέτρα, τα οποία είναι στην κατηγορία των μεγάλων σκαφών και ένα 25 πάνω δηλαδή από 24. Επίσης όσον αφορά τις, τον εξοπλισμό και τα βίντεο, τις τροχαλίες που έχουμε στις στράτες αυτές. Είναι και θέμα αρχικής, αν θέλετε, κατασκευής. Πρόκειται για σκάφη τα οποία, στα οποία τοποθετείται η κάμερα και το σύστημα παρακολούθησης ε, ανάλογα με την ε, δομή του. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου και ελπίζουμε να το συνεχίσουμε για ακόμα δύο ή τρία χρόνια. Η τεχνολογία μας επιτρέπει κάποιους ρυθμούς, δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Έχουμε προοδεύσει παρόλα αυτά. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχουμε αυτές τις ε, δυνατότητες στην διαλογή σας έδειξα αυτές τις εικόνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή συλλέγονται και αναλύονται και γίνεται η ανάλυση από τον αλγόριθμο στο Ινστιτούτο, στο Πανεπιστήμιο. Το επόμενο βήμα είναι αυτό να γίνεται επιτόπου με ένα λογισμικό επιτόπου. Επαναλαμβάνω ότι η τεχνολογία προοδεύει και μας επιτρέπει κάποιες ε, δυνατότητες που δεν είχαμε. Αν κοιτάξουμε τη σύγκριση των δικών μας στοιχείων, των ευρωπαϊκών, αυτά που έχουμε δηλαδή από το πείραμα στην Ολλανδία, με τα στοιχεία που μπορούμε να συγκρίνουμε με την Νορβηγία ή τη Νέα Ζηλανδία, διαπιστώνουμε ότι εμείς έχουμε πολύ πιο μεγάλο φάσμα αλλιευμάτων. Δεν θέλω να πω ότι στη Νορβηγία και στη Νέα Ζηλανδία αλλιεύονται μόνο ενός ε, είδους ε, ε, ηχθείες, αλλά η δική μας πολυμορφία σίγουρα μας οδηγεί σε πολύ περισσότερες προσπάθειες και πολύ πιο ευρύ φάσμα στοιχείων προς σύγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που αναφέρατε σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ακούσαμε επίσης και την απάντηση του κυρίου Σαβουρέ ότι πρόκειται για μία πολύ συγκεκριμένη ε, συμφωνία που υπογράφεται σε εκούσια βάση. Και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε ότι ξαφνικά όταν αυξηθούν οι ποσότητες ε, επιτρεπόμενων αλλιευμάτων εξαφανίζεται το πρόβλημα. Τώρα, το θέμα της Ισπανίας ε, θα μας το παρουσιάσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αλίας. Έχετε το λόγο. Η κυρία Αλίσια Βιγιαρουίθ Ιγλέσια. Good morning to everyone. I would like uh, to make... Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την παρουσίασή μου στα Ισπανικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου έχετε ε, απευθύνει να συμμετάσχω σε αυτήν την ακρόαση στην Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου και που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω την δική μας άποψη όσον αφορά τις προκλήσεις ε, του νέου συστήματος ελέγχου που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματικό, αλλά όχι μόνο. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να ε, κάνω την παρουσίαση αυτή εκ μια μιας χώρας μέλους για την οποία ε, ε, ο ρόλος της αλίας και η συμβολή ε, στην οικονομική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και επίσης γιατί η αλληλεία στην χώρα μου την Ισπανία είναι απολύτως συνειφασμένη με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα και θέλουμε να παραμείνει αυτό και στο μέλλον. Στην παρέμβασή μου, η οποία βεβαίως θα είναι σύντομη, και ενδεχομένω ε, θα μπορούσα να πω μερικά πράγματα παραπάνω στα σχόλια, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, στο γεγονός ότι η Ισπανία είναι μία από τις κεντρικέ ε, κύριε χώρες, είναι η χώρα η πιο σημαντική ε, εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεω όσον αφορά την ελιευτική δραστηριότητα και επίσης θα αναφερθώ στα προγράμματα ελέγχου και πώ εφαρμόζονται στην Ισπανία. Επίση, θα αναφερθώ και στο κοινοτικό και το διεθνές πλαίσιο και το πώς αυτά έχουν εξελιχθεί όσον αφορά το, την κοινοτική αλληλεία, έτσι ώστε να φτάσω και σε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πιο σημαντικά, καθώς επίσης και για τις ελλείψεις που έχουμε ε, διαπιστώσει στον νέο κανονισμό ελέγχου. Θα ολοκληρώσω δε εκφράζοντας κάποια συμπεράσματα και κάποιες γενικές σκέψεις. Πράγματι, η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα μέλη της της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, τον αριθμό αλλιευτικών σκαφών, ένα πέμπτο των σκαφών και των ε, αλλιευμάτων ε, και συμβάλλει στην δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας ε, και στην υδατοκαλλιέργεια και στην εξαγωγική αλληλεία αλλά και στην, με αυτές συνειφασμένη βιομηχανία μεταποιητική κλπ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές θέσεις, 20.000 περίπου θέσεις εργασίας ε, από την αρχή μέχρι το τέλος της αλλιευτικής αλυσίδας, δηλαδή από τη στιγμή της αλλιεύσης μέχρι τη στιγμή της ε, κονσερβοποίησης και της μεταποίησης. Ε, όσον αφορά την κατανάλωση και η κατανάλωση ακριβώς ενισχύει τα όσα είπα μέχρι τώρα, όπως άλλωστε ενισχύεται, ενισχύονται τα λόγια μου και από τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε και όσον αφορά αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ε, σε σχέση με όλες τις χώρες από τις οποίες εισάγουμε ή προς τις οποίες εξάγουμε. Ε, πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία έχει ιδιαίτερη σχέση ε, με και ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για τον έλεγχο την, της παράνομη παράνομης αλίας, αλία η οποία δυστυχώς εκφεύγει όποιας, όποιου ελέγχου και όποιας ιχνηλασιμότητας. Η Ισπανία έχει υψηλά ποσοστά γιατί είναι παρούσα σε πολλές αλλιευτικές ζώνες του κόσμου, ε, σε όλους τους ωκεανούς ε, της ε, Ιφιλίου και έχει μεγάλη διαφοροποίηση αλλιευμάτων και ειδών σε μερικές περιπτώσεις δε και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε σχέση δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα ψηλά όπως βλέπετε και στην διαφάνεια. Ε, στην ε, Ισπανία επί δεκαετίες έχουμε και ένα ισχυρό σύστημα επιτήρησης ε, και ελέγχου. Έχουμε το Centro de Πεσκέρο, Pesquero καθώς επίσης και την παρακολούθηση όσον αφορά την παράνομη αλία. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτό το κέντρο επιτήρησης αλίας, αλίας 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο γνωρίζουμε μέσω του συστήματος αυτού όλα τα σκάφη που βρίσκονται και με ποιο τρόπο επιχειρούν. Ε, και σε σχέση με 2.000 ε, περίπου ε, σκάφη. Μιλάμε για σκάφη πάνω από 15 μέτρα. Όσον αφορά την άναρχη παράνομη αλληλεία, πρέπει να πω ότι είμαστε σκαπανείς όσον αφορά την δημιουργία νομοθετικών κειμένων τα οποία οδηγούν εις την δίωξη αυτών των παραβάσεων και κολασίμων πράξεων. Ε, όσον αφορά δε τις περιφερειακές οργανώσεις ε, ε, αλληλείας και με αυτές συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά πολύ καλά αποτελέσματα. Ας πούμε οι Sparrow Operations, έτσι είναι γνωστές αυτές οι επιχειρήσεις, καθώς επίσης και συνεργασίες με RFMOs κλπ, Λατινική Αμερική κλπ έχουν δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα θα αναφερθώ τώρα στο πώς έχει τροποποιηθεί ε, το διεθνές περιβάλλον ε, με αναπτυσσόμενο τρόπο, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Η παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει και την αλληλεία, καθώς επίσης ε, και το γεγονός ότι έχουμε ξένες ξένους στόλους που ψαρεύουν παντού, που δεν ενδιαφέρονται όμως οι στόλοι αυτοί για την αρχή της βιωσιμότητας που όμως εφαρμόζεται και επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναφερόμαστε σε διεθνή διακυβέρνηση των ε, ωκεανών με πολλές και ενδιαφέρουσες ε, ε, προσπάθειες οι οποίες άλλες έχουν ολοκληρωθεί ή ε, ε, εφαρμοστεί, άλλες όχι. Μιλάμε για, διευρύ, για συζητήσεις και συμφωνίες οι οποίες όμως είναι ανομοιογενείς και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για διάφορες δράσεις οι οποίες όμως δεν είναι συντονισμένες και δεν είναι καθόλου διασυνδεδεμένες μεταξύ τους τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο δεν είναι δυνατόν να λείπουν από αυτόν τον ε, ε, ε συντονισμό που πρέπει να επιτευχθεί. Εδώ και χρόνια μέσω της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής, ε, μέσω ε, και της διαχείρισης επιτυγχάνουμε την βιωσιμότητα, βιωσιμότητα κυρίως περιβαλλοντική, αποφεύγοντα αποφεύγοντας τον αποδεκατισμό των αλλιευτικών αποθεμάτων κλπ. Όμως, για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε όσο γίνεται πιο καλά, ε, πλούσια και αποτελεσματικά στοιχεία. Ε, για να έχουμε, ε, πρέπει να έχουμε τα δεδομένα για κάθε παρτίδα που θα είναι σωστά και τα στοιχεία των δηλώσεων θα είναι σωστά. Δυστυχώς πολύ συχνά κατά την άποψή μου έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιστημονικά κείμενα τα οποία διήστανται μεταξύ μεταξύ και δημιουργούν ε, μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την ε, διαχείριση ε, της Αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως χαιρετίζουμε την όποια προσπάθεια των οργανισμών να δώσουν περισσότερα στοιχεία, να είναι δηλαδή σε θέση να δώσουν περισσότερα δεδομένα. Γι' αυτό χαιρετίζουμε λοιπόν, λέω, όλα τα θέματα αυτά, όπως καλωσορίζουμε και άλλα θέματα, όπως είναι ε, ο έλεγχος, όπως είναι η ε, ε, γνώση όσον αφορά την μόλυνση από πλαστικά, μικροπλαστικά κλπ. Η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα όμως έχουν περάσει λίγο περισσότερο απαρατήρητα ως στοιχεία. Νομίζω ότι θα πρέπει τα στοιχεία αυτά στον κανονισμό ελέγχου να τα αντιμετωπίσουμε. Κυρίως την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργώντα δημιουργώντας ένα level playing field ε, για όλους ε, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός αποτελεσματικός έλεγχος ε, όλων των αλλιευμάτων καθώς επίσης και να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά συστάσεις ε, ε, οι οποίες ε, ακούγονται σε διάφορα φόρα σχετικά με τη διευθέτηση της παράνομης αλληλείας και σε σχέση φυσικά και με το θέμα της ασφάλειας επί των σκαφών. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να τα λύσουμε στο μέλλον. Αυτές οι αλλαγές και στο κοινοτικό πλαίσιο θα πρέπει οπωσδήποτε να βασιστούν στο, σε σχήματα ευρωπαϊκού ελέγχου και ε, να εφαρμοστούν στην αλληλεία από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από την αλλίευση μέχρι τη μεταποίηση του ελευτικού προϊόντος. Θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τεχνολογίες πληροφόρησης ή άλλες. Έχουμε επίσης ε, και την ε, ΕΦΚΑ η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στο να βρούμε λύσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε σαφείς στόχους, σαφείς αρχές. Θα πρέπει να υπάρχει σωστό συντονισμός και συνοχή, συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων πολιτικών τη Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα στοιχεία ε, και σε όλες τις ε, εκφάνσεις. Κυρίως αναφέρομαι εις, την, εις τις κυρώσεις, καθώς επίσης και στις διευθετήσεις που αφορούν τις εισαγωγές. Επίσης θέματα όπως είναι η ερασιτεχνική αλληλεία θα πρέπει να εναρμονιστεί. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ίδιους ε, οι ίδιες προϋποθέσεις για όλους, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Όσον αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις μπορώ να πω το εξή. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι προτάσεις να είναι συνεκτικές με τις ανάγκες του τομέα. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε εφικτές και εφαρμόσιμες αρχές. Οι κανόνες, αν δεν είναι, μπορούν να εφαρμοστούν, δεν έχουν καμία έννοια. Θα πρέπει να δημιουργηθούν, ε, ας πούμε, συσχετισμοί και με την δυνατότητα, με την δύναμη μάλλον την των κινητήρων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε συνέργειες ανάμεσα στι ε, ενωσιακές πολιτικές ε, και τα εργαλεία. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην, στο, στην υλοποιησιμότητα και στην στον έλεγχο. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον ευημερία και σταθερότητα και ελπίζουμε ότι ε, σε αυτό θα συμβάλλει και ένα ικανοποιητικό αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, συνεχίσουμε, πριν φύγετε, πριν φύγετε, α, φύγατε ήδη όμως. Πριν περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, Ακούσαμε ότι η Ισπανία έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο. Ε, έχει όμως και το ρεκόρ όσον αφορά τις καταγεγραμμένες παραβάσεις. Τώρα θα εφαρμοστεί ένα αυστηρότερο σύστημα ελέγχου ε, αυτό που σημαίνει ότι θα ε, υπάρξουν λιγό, θα υπάρξει μικρότερο σχετισμός ε, των καταγεγραμμένων παραβάσεων Ισπανίας σε σχέση με άλλων χωρών. Είναι σωστή η σκέψη μου. Ναι, το ε, είπα και στην παρουσίαση. Η εξέλιξη στα συστήματα των συστημάτων ελέγχου στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, τα 20 μάλιστα τελευταία χρόνια, τότε που άρχισε να λειτουργεί ε, το ε, κέντρο παρακολούθησης της αλίας, είχαμε πολύ θετικές εξελίξεις, γιατί κάθε φορά, όλο και περισσότερο δηλαδή, μπορούσαμε να ελέγχουμε του, τα αλλιευτικά σκάφη μεγάλα και ε, μικρότερα. Πιστεύω ότι ε, χρειάζεται οπωσδήποτε ε, μια σημαντική επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, σε χρηματικούς, οικονομικούς πόρους. Εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια, έστω και αν ήταν δύσκολη. Έχουμε λοιπόν σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση του, της, ε, των ελευθερικών σκαφών στις παράκτιες περιοχές αλλά ε, και ε, οπουδήποτε αλλού. Το έλεγε προηγουμένως και η κυρία Αγγιλέρα Μπορεί να υπάρξουν πολλές ε, ε, παραβάσεις. Έχουμε ε, μεγάλες περιπτώσεις απάτης ας πούμε, και παραβάσεων στη διάρκεια του χρόνου, αλλά έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει συσχετισμός. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν νέες ομάδες, όπως έγινε ας πούμε για την επιτήρηση της παράνομης άνεργης αλληλείας. Θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες έρευνας, διαρεύνησης των απατών ή οποιονδήποτε αδικημάτων σε σχέση με την ε, ε, αλίευση και πιστεύω ότι διαρκώς θα βελτιώνεται το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Τεχέρα από την ε, Ισπανική Οργάνωση Ελιέων. That picture shows just exactly what I feel about Brexit. Ε, αυτή η εικόνα πραγματικά δείχνει τον τρόπο τον οποίο αισθάνομαι για τον Brexit. Bueno. <clears throat> Buenos Καλημέρα, bon día σε όλους. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να στείλω να στείλω ε, τι τον χαιρετισμό μου στην οικογένεια του Εντιβίνα Παστόρα, γιατί η οικογένεια ε, της ε, Αλίας στην Γαλλικία έχασε ένα μέλος της και λυπούμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που, μας, που με καλέσατε σε αυτήν την ακρόαση. Είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό το ότι μπορώ να είμαι σήμερα εδώ έτσι ώστε να ακούσετε πραγματικά την άποψή εγώ είμαι γενικός ε, γραμματέας σε μια οργάνωση πλειοκτητών. Ε, είμαι ε, εκ των σπουδών μου δικηγόρος ε, αλλά ε, το σημαντικό είναι ότι εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αλία και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να περνάς ώρες πάνω σε ένα λιευτικό σκάφος. Εγώ εδώ δεν είμαι ούτε για να εκπροσωπήσω λόμπι, ούτε για να εκπροσωπήσω ομάδα ε, συμφερόντων. Εγώ δεν έχω καμία ανάγκη να το κάνω και δεν έχω κανένα λόγο να αλλοιώσω την πραγματικότητα απέναντί σας, ούτε και θέλω να στρεβλώσω την κατάσταση κατάσταση ε, ε, πραγματικά δεν χρειάζομαι καθόλου να χειραγωγήσω την κοινή γνώμη. Θέλω μόνο να ακούσετε από μένα την πραγματικότητα της αλίας. Αυτό και τίποτα άλλο. Δεν θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες γιατί σε 10 λεπτά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα έπρεπε να τροποποιηθεί στο έγγραφο που υποβάλλει η Κομισιόν. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτό το έγγραφο ε, και ότι εδώ, εδώ σας δείχνω δείχνω πραγματικά αυτούς τους δύο ανθρώπους, ο ένας ε, δείχνει να είναι σε πανικό και ο άλλος σε μεγάλη θλίψη. Αυτή είναι η κατάσταση της αλίας σήμερα ε, και ε, πραγματικά, πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε πλέον απέναντί μας έναν κανονισμό ο οποίος θα είναι πιο λογικός και πιο εφαρμόσιμος. Πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ σας διαβάζω, σας δείχνω μάλλον αυτό που γράφτηκε στον τύπο της ε, Γαλλία, ε, Γαλλικίας ε, ότι η ΕΦΚΑ έχει αυξήσει τις επιθεωρήσεις κατά 30% αλλά φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι περιπτώσεις απάτης. Θα... Να σας πω το εξής. Εγώ προέρχομαι από την Λακορούνια, είναι ένα πολύ σημαντικό αλλιευτικό λιμάνι και να σας πω ότι είχαμε περίπου 240 επιθεωρήσεις από την αρχή του χρόνου. Ε, ένας και ε, ένας από τους ε, ε, μεγαλύτερους στόλους με απλάδια είχαν αυτές, αυτούς τους 240 ελέγχους με 15 διαδικασίες παράβασης. Μονάχα 10 αφορούν ακριβώς την, τον έλεγχο. Είναι οι υπόλοιπε 5 έμεσες γιατί δεν έχουν σεβαστεί ας πούμε το ποσοστό της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 Εάν υπάρχουν τόσο λίγες παραβάσεις, ε, ε, ε, ίσως σημαίνει ότι στην Ισπανία έχουμε την Guardia Civil της θάλασσας, έχουμε επιθεωρήσεις από τις αυτόνομες περιφάρειες και επιθεωρήσεις από την Κεντρική Αρχή που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο να ξεφύγει κανείς από αυτές τις επιχειρήσεις. Και διαφορετικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ πανούργοι οι ψαράδες και ξεφεύγουν, ξεγλιστράνε. Ε, αλλά νομίζω ότι ε, μπορούμε όμως, αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, να πούμε ότι είναι ε, τίμοι οι, ε, οι, οι ψαράδες και δεν κάνουν απάτες αυτή, να σας πω, η ε, πρωτοβουλία από που ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε, όταν είχαμε το feedback, λίγες ε, ήταν ε, οι οργανώσεις οι οποίες ανταποκρίθηκαν και όταν μπήκε σε διαβούλευση το 2018, έξι μονάχα οργανώσεις ευρωπαϊκές απάντησαν σε αυτήν την διαβούλευση. τι λέει η Κομισιόν όσον αφορά την ε, εφαρμογή ε, του παρόντος ε, κανονισμού λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν καλύψει τις κύριες δραστηριότητες ελέγχου και έχουν, έχουν θεσπίσει τα όργανα τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και την επιτήρηση των λευτικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ θα πρέπει όμως να διαπιστώσουμε ε, ότι ε, η Κομισιόν οπωσδήποτε λέει ότι κάποιες χώρες δεν εφαρμόζουν καλά τον κανονισμό. Ε, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πάνω στα θέματα αυτά, γιατί ήδη η Κομισιόν έχει αναφερθεί στα προβλήματα. Το έγγραφο της Κομισιόν στην ουσία είναι υποχώρηση. Και αυτό θέλω να το θυμάστε, το λέω σαν σλόγγαν δίνει στην ε, Κομισιόν αύξηση της ε, δυνατότητας ε, να νομοθετήσει σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και επίσης δεν υπάρχει καθόλου κριτική από την ε, Κομισιόν, ε, γιατί υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικότητας λέμε. Οκ, αλλά μήπως αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ε, ανάμεσα στην πραγματικότητα ε, και τους ελέγχους. Τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα και νομίζω ότι εδώ γίνεται περίπλοκος ο νέος κανονισμός βάζοντας πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες είναι ανώφελες. Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη της η Κομισιόν και όλοι οι υπεύθυνοι. Κάτι πάρα πολύ πολύ ε, σαφές. Ε, δηλαδή ότι η αλληλευτική δραστηριότητα είναι δύσκολη και περίπλοκη και επικίνδυνη ε, και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε το πλήρωμα να αφιερώνεται 100% στην προστασία της αλληλευτικής τους δραστηριότητας αλλά και στην προστασία της ίδιας τους της ζωής. Θα πρέπει οπωσδήποτε το πλήρωμα να οργανωθεί σωστά και θα πρέπει το πλήρωμα να μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ αντίξωες συνθήκες. Πού βρισκόμαστε όμως τώρα. Βρισκόμαστε στο εξή. Όταν κάνει η Κομισιόν ε, ε, ερωτήσεις και απαντήσεις λέει ε, ότι θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό και σε απλούστευση. Αλλά αυτό δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο τι είναι, δηλαδή με, το, με τον Big Brother, με, τα μάτια του μεγάλου αδερφού ε, θα παρακολουθεί ας πούμε όλους τους ε, ε, ψαράδες και αυτό θα δώσει καλά αποτελέσματα και θα γίνει η πιο αποτελεσματική ε, επιτήρηση. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θα πρέπει πραγματικά να προστατέψει τους αλληλείς και στην δραστηριότητά τους και στην ασφάλειά τους. Αλλά ε, τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Ε, βρίσκεται το ότι η Κομισιόν μας λέει ότι το σύστημα ελέγχου και της εφαρμογής ε, θα είναι καλό και για την φήμη, την καλή φήμη του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πραγματικά δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο να το ακούμε αυτό, ότι δήθεν ε, η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζεται και διακυβεύεται από την ε, αλία. Η αλία είναι πραγματικά μια οικονομική δραστηριότητα. Είναι μια δραστηριότητα που αφορά την υγεία, γιατί δύο φορές ψάρι την εβδομάδα είναι η καλύτερη δίαιτα, αν όχι παραπάνω. Επίσης, το, ο συσχετισμός της θάλασσας και της αλίας με τη διατήρηση των ποσοστών οξυγόνου. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουν πει όλοι οι επιστήμονες. Τώρα, ε, ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει ε, να αλλάξουν. Όλες οι δραστηριότητες ε, και κομισιόν δεν είναι ίδιες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια διακυβέρνηση αποκεντρωμένη. Θα πρέπει να αποφύγουμε υπερβολική σχετικά βαριά ε, κανονιστική ρύθμιση η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στην ε, ε, διοίκηση αλλά θα, θα, θα είναι και δύσκολη στην εφαρμογή. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε την θέση που τους αρμόζει σε, αυτές, σε αυτά τα συμβουλευτικά όργανα, συμβούλια. Πραγματικά θα, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να δείτε λίγο ποια είναι η δουλειά που έχει κάνει αυτό το ε, συμβουλευτικό Συμβούλιο ε, μέσα από την, από το ψήφισμά του, μάλλον την έκθεσή του υπαριθμών 127 της 13ης Μαρτίου του 2019 για να καταλάβετε πραγματικά ε, πώς έχουν τα πράγματα. Ε, θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας το εξής, κάτι που δεν θέλω να ξεχάσετε. Ο έλεγχος δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός. Ε, βεβαίως είναι θεμελιώδες στοιχείο για την βιώσιμη αλληλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρακαλώ να θυμάστε όταν νομοθετείτε ότι ε, θα πρέπει να, σκεφτώ, να σκεφτόσαστε και τα ψάρια αλλά και τους ψαράδες. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much indeed. And uh, Mr. Acheta, the Vice President of uh, <laughs> Federico Pesca from Italy. Ο κύριος Ατσέτα από το Feder Pesca της Ιταλίας. Ξέρω ότι η γραμματεία εδώ γελάει γιατί η προφορά μου ήταν πάρα πολύ αστεία. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μου δίνετε το λόγο. Ζητώ ε, συγγνώμη που ε, έκλεισε η φωνή μου γιατί κάνει κρύο εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν το περίμενα αυτό. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε ε, να ε, σας μιλήσω για, κάποιες, ε, για κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αλληλείς και σε σχέση βεβαίως και με τον νέο κανονισμό για τον έλεγχο. Η πρώτη έννοια που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην αλληλεία μεγάλης κλίμακος και μικρής κλίμακος, δηλαδή για σκάφη πάνω ή κάτω από 12 μέτρα. Όταν μιλάμε για σκάφη κάτω των 12 μέτρων, ε, γίνεται, ε, αναφερόμαστε και στα σκάφη ε, της ε, των ερασιτεχνικών, ε, τις ερασιτεχνικές μορφές ε, αλίας, αλία με καλάμι, καθώς επίσης και αλία με παραγάδια. Κατα... Κατανοώ βεβαίω του λόγου για του οποίου οδηγήθηκε η Κομισιόν ε, να συγγράψει και να υποβάλει αυτόν τον ε, κανονισμό έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο έλεγχο. Παρ' όλα αυτά όμω δεν μπορώ να ξεχάσω ότι κάποια άρθρα φαίνεται να. Ε, να λένε ότι τελικά η αλληλεία αναψυχής ε, είναι αυτή η οποία εκφεύγει του συστήματος ε, ελέγχου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε και να προσαρμόσουμε τις ε, υποχρεώσεις ελέγχου σε δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Όταν μιλάμε για σκάφη κάτω των 12 μέτρων αναφερόμαστε και σε πολλά σκάφη τα οποία κάνουν, ε, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα συστήματα. Ε, έχουμε δηλαδή, όπως σας έλεγα, τα ε, παραγάδια, τα παρασυρώμενα πλάδια. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν μονάχα την μικρής κλίμακος αλία. Ε, ε, επίσης, ε, κάτω των 12 μέτρων έχουμε πάρα πολλά σκάφη τα οποία δεν έχουν καν κινητήρα. Μιλάμε για μικρά σκάφη τα οποία δουλεύουν μόνο χειροκίνητα με δίκτυα. Και αυτή είναι η ιταλική πραγματικότητα τουλάχιστον. Τα σκάφη αυτά ε, αντιπροσωπεύουν ακριβώς την ιστορία. Είναι το πρόσωπο, αν θέλετε, της ε, ε, μικρής αλίας, της παράκτιας αλίας των κρατών μας. Αυτά τα σκάφη θα πρέπει οπωσδήποτε να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε έλεγχο, αν μη τι άλλο, λόγω του πολύ χαμηλού αλλιεύματος στους ε, κανονισμούς ε, φαίνεται ότι συχνά ε, παρανοείται ή παραβλέπεται η ιδιαίτερη κατάσταση του τομέα. Αυτό που ονομάζουμε επίσης και με συμβρινοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι έχουν τα τελευταία χρόνια δημιουργηθεί, θεσπιστεί κανονισμοί ε, οι οποίοι πραγματικά δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στους μικρούς ερασιτέχνες ε, αλληλείς. Και τούτη η πρόταση κανονισμού, κύριε Πρόεδρε, στην ουσία θέλει να αποθαρρύνει την παρανομία. Αλλά εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ε, εδαφικές ιδιαιτερότητες, διατρέχουμε τον κίνδυνο να αυξηθεί αυτή η παραβατικότητα. Έχω εδώ φέρει μερικές πολύ λίγες διαφάνειες οι οποίες αναλύουν κάποια άρθρα ε, της προτάσεως. Ξεκινώ όμως από μία παρατήρηση. Ε, η ε, εραστεχνική αλληλεία δεν είναι το απόλυτο κακό και επομένως θα πρέπει να προστατευτεί ε, και όχι ε, να χτυπηθεί ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέγεθος και επομένως να προβλεφθούν κάποιες εξαιρέσεις. Εξ αρχής θέλω να πω ότι ε, οπωσδήποτε δεν θέλουμε να μην ελέγχεται αυτή η μορφή αλίας. Όχι, εμείς αντιθέτως λέμε ότι θα πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα εφαρμόσιμα μέτρα, τα οποία όμως θα είναι λογικά και εφαρμόσιμα για τα μικρού μεγέθους σκάφη, γιατί διαφορετικά ε, αυτά τα μικρά αλλιευτικά σκάφη θα μπορούσαν να ε, ε, δημιουργήσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και να είναι κατά κάποιο κάποιο τρόπο μπροστάριδε, αυτό είναι την παραβατικότητα. Αυτό θέλουμε λοιπόν να πούμε, να μην μπερδέψουμε ακόμα περισσότερο και να μην δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο τους μικρούς αλληλεί και τους ερασιτέχνες αλληλεί μας. Με, την, με τις συγκεκριμένε προτάσεις κανονισμού θέλουμε επίσης να αποφύγουμε επιπλέον επιβάρυνση των εργαζομένων. Υπάρχουν ε, ε, πραγματικά διατάξεις οι οποίε ε, δυναμητίζουν την ίδια τη δραστηριότητα όσον αφορά συγκεκριμένα το άρθρο 9 του κανονισμού όσον αφορά το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μικρά τα σκάφη έτσι ώστε να υποχρεωθούν να έχουν συστήματα εντοπισμού και ταυτοποίησης ε, στο σκάφος. Θα πρέπει οπωσδήποτε τα σκάφη πάνω από 12 μέτρα να ε, ε, ε, έχουν την υποχρέωση για τέτοια συστήματα. Ε, αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή ε, ε, κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες είχαν δοθεί στα κράτη-μέλη με το νέο κανονισμό θέλουν να διαγραφούν. Πρόθεση είναι να διαγραφούν. Επίσης λέμε ότι κάτω από 12 μέτρα θα πρέπει να, λάβει υπό, να ληφθούν υπόψη είτε οι ιδιαιτερότητες λόγω του μήκους του σκάφους, είτε οι ιδιαιτερότητες λόγω της εδαφικότητας, λόγω της γεωγραφικής ε, θέσης. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν διατάξεις ε, οι οποίες δεν πρέπει, δεν είναι δυνατόν, πώς να σας το πω, δεν είναι δυνατόν να μπουν τέτοιες διατάξεις μέσα σε ένα ευρωπαϊκό κανονισμό. Ας ασκήσουμε την αρχή της περιφερειοποίησης ε, όσον αφορά όμως το άρθρο 14 παράγραφος 1. Στην πρόταση κανονισμού η Κομισιόν προβλέπει ε, ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταστρώματος για κάθε σκάφος. Στην παρούσα κατάσταση σκάφη πάνω από 10 μέτρα υποχρεούνται να έχουν τέτοιου είδους ε, ημερολόγια καταστρώματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις που έκανα πριν και λαμβάνοντας υπο... για, τα... Ε, για την αριστεχνική ε, αλία και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε σε αυτήν την περίπτωση αλίες που είναι πιο ηλικιωμένη, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις για γέρους με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στους νεότερους, άρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και λέω ότι για να αποφύγουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες ε, ε, ε, δεν θα πρέπει οι μικροί μας αλληλείς να υφίστανται τέτοιες κυρώσεις. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει λογικά να ε, ε, εξαιρεθούν αυτές, αυτά τα σκάφη τα οποία δεν χρειάζεται να κρατούν τέτοιου είδους καταγραφές εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις οι οποίες ήδη υφίστανται όσον αφορά συγκεκριμένα είδη όπως ας πούμε είναι οξυφίας. αλλιεύματα κάτω από τα 50 ε, κιλά δεν θα χρειάζεται να καταγράφονται ε, και θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα ανοχής 10% στις ε, εκφορτώσεις, λέει η παράγραφος 4. Εμείς θα μπορούσαμε να μειώσουμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 30 ή 40 κιλά πριν αρχίσει η εφαρμογή των κυρώσεων. Αυτό θα βοηθούσε. Για σκεφτείτε λίγο. Ε, πολύ μικρές ε, παρτίδες, 2-3 κιλών, μισού κιλού ε, που θα πρέπει να δηλώνονται στην εκφόρτωση από σκάφη τα οποία είναι κάτω από 10 μέτρα. Αλλά εάν μιλήσουμε για 50 κιλά τότε δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 για την ε, ηλεκτρονική υποβολή του logbook, η Κομισιόν ε, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν μονάχα δύο κατηγορίες, ε, κάτω από 12 και πάνω από 12. Εμείς θα προτείναμε να υπάρχει μονάχα μία κατηγορία κάτω από 12 ε, μέτρα καθαρό ε, μήκος ε, και μετάδοση των δεδομένων μία φορά την ημέρα. Ακόμα και για αυτούς που έχουν έξοδο αλλιευτική πάνω από μία μέρα. Ε, και επίσης μονάχα στην επιστροφή στο λιμάνι ε, θα πρέπει να καταγράφονται τα δεδομένα. Εγώ και ε, αυτό 24 ώρες από την αναχώρηση από το λιμάνι. Όμως, το άρθρο 17 είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εάν δεν ε, ελεγχθεί και θεωρηθεί σωστά θα μας προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες. Ε, αυτή τη στιγμή ε, έχουμε υποχρέωση πρώτερη κοινοποίηση για την Πελούγα και για τον Ξηφία. Κάθε χώρα μέλος έχει την υποχρέωση διακόπτει ο μιλητή. Εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε την ιδέα, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, για τα σκάφη πάνω από 10, 10 ε, μέτρα, ε, να ε, υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε που γίνεται η ε, επιβίβαση. Ε, ε, σε πολλές περιπτώσεις δε αυτά τα σκάφη δεν έχουν καν δυνατότητα ψήξης και επομένως καταλαβαίνετε αν μιλάμε για ακόμα μικρότερα σκάφη και για ακόμα μικρότερες κλίμακας αλλήλεία, εάν αυτά τα σκάφη θα έχει υποχρέωση πρώτερης κοινοποίησης θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα πω το εξής τελειώνοντας, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές ε, για να μπορέσει κανείς να έχει καλύτερη, καλύτερο έλεγχο μπαίνει διαρκώς σε όλο και μεγαλύτερη λεπτομέρεια ε, και εκεί επιβαρύνεται εν τέλει ο πιο μικρός. Δεν είναι δυνατόν ε, βεβαίως να υπάρχει κανονισμός ο οποίος να είναι κατάλληλος για όλα τα είδη των αλλιευτικών σκαφών. Ε, επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε τα στοιχεία να είναι διαφοροποιημένα. Για τα μικρά σκάφη, για την αλληλεία αναψυχής θα πρέπει να βρεθούν ξεχωριστές υποχρεώσεις με ανάλογες ε, κυρώσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα μεταχείρισης όλων των αλλιέων σε όλα τα κράτη-μέλη. Well, thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε με αυτόν τον ε, κύκλο των ομιλητών. Επειδή θέλω να έχει και η Επιτροπή αρκετό χρόνο στη διάθεσή της για να παρέμβει, θα ήθελα οι παρεμβάσεις να παραμένουν κάπου το ένα λεπτό. Η κυρία Αγγιλέα λοιπόν έχει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. <clears throat> Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές ε, για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπαν. Νομίζω ότι όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι ήταν όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Μας βοηθούν καλύτερα να <laughs> καταλάβουμε την πραγματικότητα. Οι δύο τελευταίες ε, παρεμβάσεις ε, που εκπροσωπούσαν τους κλάδους ε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η τελευταία που μίλησε για την ερασιτεχνική αλληλεία. Ναι, είναι πραγματικά, δεν είναι δυνατόν ανώμια πράγματα να τα βάλουμε στο ίδιο σακί και να τα ελέγχουμε με τον ίδιο όμοιο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Ένα πράγμα είναι βεβαίως το ότι μιλάμε για ε, στόλο ανώμιο όσον αφορά και το, τις δυνατότητες ε, και το μέγεθος και επομένως δεν είναι δυνατόν ε, να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά να ελέγχονται φυσικά. Γρήγορες ερωτήσεις αν είναι δυνατόν, όχι πολλά σχόλια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εντάξει, θα μπω στο ψητό λοιπόν. θα ήθελα να ρωτήσω τους δύο τελευταίους εισηγητές. Όποιος θέλει να απαντήσει. Ποια μεθοδολογία, ποιες μεθόδους μπορούμε να εισάγουμε έτσι ώστε κάθε μορφή αλίας και η να ε, ενταχθεί σε ένα ε, λογικό σύστημα ελέγχου. Κατά τη δική τους άποψη. Επόμενος ομιλητής ε, κύριος Μιγιάν μόνο. Ευχαριστώ πολύ τις ε, τρεις, ε, τους τρεις παρεμβαίνοντες. Θα ήθελα όμως ε, κυρίως να αναφερθώ στον Ιταλό ομιλητή Την διαφοροποίηση της ερασιτεχνικής αλίας από άλλες μορφές αλίας. Είναι λογικό. Είναι πολύ σημαντική η ερασιτεχνική αλία, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και γιατί λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ε, τον παραδοσιακό ε, χαρακτήρα, τις ε, λίγες ώρες αλίευσης, τις λίγες ώρες που βρίσκεται κανείς στο σκάφος και στη θάλασσα, θα πρέπει να βρεθούν κάποιες, κάποιοι ειδικοί τρόποι, γιατί αυτά τα οποία προτείνονται είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικά και μπορεί να ο κύριος στόχος να είναι ε, ο έλεγχος, αλλά αυτό, πρώτερη, ε, ανα, πρώτερη ανακοίνωση, πρώτερη κοινοποίηση, ε, ηλεκτρονικό logbook, ε, υπολογισμός της εκφόρτωσης, το να άλλο. Ε, όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να ε, τα βάλουμε στην πλάτη των ερασιτεχνών ψαράδων. Η ερασιτεχνική αλία πραγματικά πρέπει να ελέγχεται, αλλά θα πρέπει να δώσουμε κάποια ειδικά στοιχεία όσον αφορά αυτή τη μορφή και συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο κύριος Ατσέτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα έχει να κάνει με το εξή. Γνωρίζουμε ότι η Μεσόγειος είναι η θάλασσα εκείνη ε, στην οποία λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη παραλίευση και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις χώρες της ε, ε, Βόρειας Αφρικής αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι αριθμοί μικρής κλίμακα αλευτικών σκαφών και αλλιών που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στη μείωση της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο. Για παράδειγμα, το να ε, ε, εφαρμοστεί, να επιβληθεί η τήρηση ενός ε, ημερολογίου σκάφους δεν θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν έχουμε και πολλές ανάλλακτικές. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Τώρα το δεύτερο ερώτημα προς την Επιτροπή. η Επιτροπή σε πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού ελέγχου έχει προτείνει την αναδιατύπωση ε, των διατάξεων 59, 60 και 64 σε ό,τι αφορά δηλαδή τη στάθμιση, το ζήγισμα δηλαδή των ε, λευμάτων κατά την εκφόρτωση. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι αλληλείς έχουν δαπανίσει χιλιάδες ευρώ έτσι ώστε να έχουν εξοπλισμό ακριβώς για να λαμβάνει η χώρα η ζήγηση εν πλώ πάνω στο σκάφος. Τι θα κάνουν λοιπόν με όλο αυτό το εξοπλισμό που αγόρασαν οι αλληλείς. Κυρία Κόντε, τώρα έχει το λόγο, Α, όχι, η κυρία Μάμερ πρώτα. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενημερωτική η σημερινή παρουσίαση ε, από τον κύριο Πασχάλ και ιδιαίτερα ο Ιταλός ε, ε, κύριος και ο Ισπανός ε, κύριος. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ε, ακούσαμε δεν ξέρω προς ε, ποιον να απευθύνω την δική μου ερώτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι η τεχνολογία στην οποία αναφέρεστε ε, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μόνο αυτή την ε, περίοδο έχει αρχίσει να εξετάζεται ένα δυνητικό σύστημα για την επιβολή ελέγχων. Ε, πού βρισκόταν λοιπόν όλα αυτά τα συστήματα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την καταστροφή των αποθεμάτων στην στα, δυτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ό,τι αφορά την ε, ε, αλληλεία που λαμβάνει η χώρα με, ηλεκτρικά, με ηλεκτρισμό, γιατί δεν εφαρμόζονται τώρα, ε, δεν εφαρμόζονταν μέχρι τότε αυτή η έλεγχη. Ε, λοιπόν ε, μέτρα τα οποία θα επιβάλλουμε ε, θα πρέπει να τεσταριστούν πρώτα για επί σειρά μηνών και να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αλλιέων και όχι στις ανάγκες των ελεκτικών αρχών και θα ήθελα να σας προτείνω να έχουμε αλληλεί από κάθε κράτος μέλου, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στι συνεδριάσει μας ανά τρίμηνο. Ευχαριστώ κύριε Σίτηρη. Ευχαριστώ λέει ο Ε, Κύριε Κόντε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένας από τους στόχους του κανονισμού ελέγχου είναι να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο των ελέγχων και να εγγυηθεί την σωστή εφαρμογή από όλες τις χώρες. Ε, εγώ περίμενα να ακούσω όλες τις παρεμβάσεις και μετά να πάρω το λόγο. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε και πρέπει να πω ε, ακούσαμε και καινοτόμα έτσι, στοιχεία επιστημονικά. Αλλά εγώ προέρχομαι από το Βένετο, όπου ε, ε, έχουμε πραγματικά τις μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην, του αλληλευτικού τομέα και τους μεγαλύτερους τόλους. Ε, νομίζω ότι δεν έχει ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, ε, δεν έχουν ληφθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ε, της αλίας στη Μεσόγειο. Σίγουρα μιλάμε για σκάφη τα οποία δεν είναι καθόλου 20 και 40 μέτρα. και όλα αυτά τα νέα στοιχεία, οι κάμερες στα σκάφη, το ηλεκτρονικό logboard και τα logbook και τα λοιπά, σημαίνει κόστος μεγάλο. Η συζήτηση που ξεκίνησε τον Ιούλιο στην Κομισιόν, ε, το Ταμείο Αλίας και Θαλάσσης ε, είχε πει ότι θα δώσει κάποιους πόρους ε, για την αγορά αυτών των εξοπλισμών στους μικρούς αλίες. Θα δώσει το ΦΕΑΜΠ αυτά τα χρήματα, ρωτώ την Κομισιόν. Επίσης έχουν προβλεφθεί ε, κάποιοι πόροι για κατάρτιση έτσι ώστε ε, να ληφθούν υπόψη και αυτοί οι αλληλείς που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Σατσέτα. Επίσης, ε, τι γίνεται με αυτό που είπε ο κ. Σατσέτα προηγουμένως, δηλαδή να μην χρειάζεται ηλεκτρονικό βιβλίο καταστρώματος για τα πλοία κάτω από 10 μέτρα. Uh, Ευχαριστώ. Ε, οι μιλητέ μα, οι πάνελιστ, δηλαδή, αν έχουν να θέσουν κάποια ε, δικά του ερωτήματα, μπορούν να το κάνουν. Ναι. Δεν υποχρεούνται να το κάνουν. Ναι, Αλλά όλοι μα θεωρούμε βέβαια προφανώ ότι οι διατάξει ε, για τα μικρότερα σκάφη θα πρέπει να είναι λίγο πιο ήπιε αλλά τι ακριβώ εννοούμε μικρά σκάφη. Δηλαδή 12 μέτρα, όταν λέμε στα 12 μέτρα ένα σκάφο είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή μπορεί να αλλιεύσει αρκετά. Ε, και από εκεί και μετά βέβαια, ε, αν δεν έχουμε ένα σύστημα παρακολούθηση των σκαφών, πώ μπορούμε να γνωρίζουμε πού ακριβώ βρισκόνται όλα αυτά τα σκάφη, πού αλλιεύουν δηλαδή. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να προβλεφθεί μια εξαίρεση σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα, δηλαδή εντοπισμού του για τα μικρά σκάφη. Ε, αλλά εντάξει, να ακούσουμε του ε, ομιλητέ, του πανελίστε δηλαδή. Πρόσωπο από την Ισπανία. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, καθώς επίσης και η γνώση των μικρών ε, σκαφών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν την δυνατότητα να δώσουν στοιχεία ε, όσον αφορά τις μικρές, ε, τα μικρά φορτία, λέει η κυρία Βιγιαουρίθε Ιγλέσιας, όσον αφορά τα, την καταγραφή των αλλιευμάτων πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, να γίνει τέτοια καταγραφή και για τα σκάφη της ε, ε, της εραστεχνικής αλίας και για τα σκάφη μικρού μεγέθους γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να γίνει και πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος μας. Όμως θα πρέπει ο έλεγχος αυτός και οι διατάξεις αυτές ε, και η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας να λάβουν υπόψη είναι τις ιδιαιτερότητες ε, του κλάδου αυτού, του τμήματος αυτού. Ε, ας πούμε έχουμε κινητά τηλέφωνα, έχουμε ε, τεχνολογία αντίστοιχη με τα smartphones και νομίζω ότι μπορούμε και στα σκάφη της αεραστεχνικής αλίας να βάλουμε κάποια τέτοια συστήματα και με τον τρόπο αυτό ε, η κατάσταση γενικής ασφάλειας για όλους όσοι λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα, οι συνθήκες λέω θα γίνουν πολύ καλύτερες. Θέλετε ξανά το λόγο, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δύο εβδομάδες, πριν από δύο εβδομάδες, εμείς κάναμε ε, monitoring, επιτήρηση με τα ε, κινητά τηλέφωνα, αλλά είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο και ούτως ή άλλως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ε, συνέχεια αυτά τα, τα, κινητά τηλέφωνα την ώρα που έρχονται τα κύματα κατά πάνω τους και την ώρα που πρέπει να κάνουν ένα σωρό πράγματα με τα χέρια τους. Μα είναι φοβερό αυτό που λέτε point made. I don't know if you wish to come back to that, but uh, I mean, ε, the point is the technology can be. Δεν ξέρω αν θέλετε να επανέλθετε σε αυτό. Η τεχνολογία μπορεί να είναι αυτή που είναι. Ο κύριο Ατσέτα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ε, η κυρία Βουλευτής μόλις τώρα. Βρισκόμαστε σε μια βάρκα, σε ένα ε, μικρό σκάφος. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εγώ άκουσα και προηγουμένως ε, την εκπρόσωπο ε, από τον εκπρόσωπο τη, της υπηρεσίας ελέγχου της αλληλείας ότι ε, κάνουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα, ξεκινάμε με τέσσερα σκάφη. Δεν κατάλαβα όμως που μπαίνουν τα μικρά σκάφη εδώ, γιατί εδώ μιλάμε ε, για ε, σκάφη κάτω από 12 μέτρα. Και εδώ πρέπει να πω ότι με μεγάλη έκπληξη αλλά και προβληματισμό ακούω διάφορα πράγματα, γιατί εμείς θα πρέπει να πάμε μετά στις χώρες μας και να μιλήσουμε, να πούμε στους ψαράδες μας τι ακούσαμε ε, και εδώ μιλάμε για την εφαρμογή ε, καμερών ακόμα και σε ε, πολύ μικρά σκάφη, γιατί διαφορετικά θα, αν δεν βάλουν τις κάμερες αυτές, θα βρίσκονται σε κατάσταση παράβασης. Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα τι γίνεται. Πώς θα γίνει να ελέγξουμε στην Μεσόγειο, ας πούμε, αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, αυτούς που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική κλπ. Κοιτάξτε, εδώ και 20 χρόνια επιβάλλουμε στους ψαράδες μας άκαμπτους κανόνες. Ε, στην ουσία τους ε, ε, αναγκάσαμε τους ανθρώπους να μην πηγαίνουν πλέον στη θάλασσα. Έχει μειωθεί κατά 50% ο στόλος, έχουν μειωθεί κατά 50% οι ψαράδες και ακόμα και τώρα Ακόμα και τώρα έχουν μειωθεί τα έσοδα ε, και ακόμα στρεφόμαστε ε, και δείχνουμε με το δάχτυλο τους ψαράδες, λες και αυτοί ευθύνονται για όλους και για τα πάντα. Δεν μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή, δεν μιλήσαμε για την ε, κατάσταση με αυτούς που έρχονται και ψαρεύουν από την Αφρική. Εμείς λέμε πρέπει να ανοίξουμε την ομπρέλα χωρίς να βρέχει, μήπως και βρέξει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι πλέον εδώ και από την υπηρεσία ελέγχου της Αλίας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να κοιτάξουμε και τις ιδιαίτερες κατηγορίες και τις ειδικέ ανάγκες όλων αυτών που είναι μικρή αλής. Είμαστε όμως σε πολύ πρώτο στάδιο ανάπτυξης αυτών των νέων συστημάτων. Το θέμα της χρηματοδότησης, παραδείγματος χάρη, ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος. Και σίγουρα όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλίας, δεν ε, έχουμε δώσει ειδική έμφαση στο θέμα της απλοποίησης και της σωστής εφαρμογής και ενιαίας εφαρμογής από όλα τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έχω σημειώσει πάρα πολλά από αυτά που άκουσα. Το θέμα του κόστους, το οποίο αναφέρατε εσείς, αλλά και πολλοί από τους παρεμβαίνοντες. Η Επιτροπή στο νέο κανονισμό, η έχει προτείνει ήδη να υπάρχει μία ειδική, αν θέλετε, πρόβλεψη και εξαίρεση για όλους αυτούς ε, οι οποίοι προβλέπουν ε, την εγκατάσταση νέων μηχανισμών, νέων τεχνολογιών για έλεγχο. Και βεβαίως θα καλυφθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ε, για το σύστημα CCTV. Εάν λοιπόν πιστεύετε ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει τέτοια κάλυψη, αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί. Το θέμα της κατάρτισης επίσης και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί το κόστος του ε, από το κανονισμό EMFF. Αυτό ήδη γίνεται, είναι όμως θέμα ε, ευθύνης και αρμοδιότητας των κρατών μελών να το υποβάλουν σαν πρόταση. Το τελευταίο κομμάτι αυτής της ακρόασης έδωσε ειδική έμφαση και προσοχή στα μικρά αλλιευτικά σκάφη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η ερασιτεχνική αλία. Δεν μιλάμε μόνο για μικρά αλλιευτικά σκάφη επαγγελματικά. Σήμερα λοιπόν στη μελέτη αντικτύπου που κάνουμε, επαναλαμβάνω ότι, και εδώ απευθύνομαι στον τελευταίο μιλητή, υπάρχει για κάτω από 50 κιλά αλλιεύματα η εξαίρεση από την υποχρέωση της α, αναφοράς και κάθε χρόνο για 350.000 τόνους, μόνο για τη Μεσόγειο βλέπετε, είναι 150.000 τόνοι, οι οποίοι τελικά περνάνε κάτω από το, την υποχρέωση αυτή. Δεν έχουμε πληροφορίες, δεν ξέρουμε γιατί αλλιεύματα αναφερόμαστε. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε και να, κυρώσουμε, και να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κανέναν, αλλά πρέπει να διαθέτουμε στοιχεία επιστημονικά αρκετά και από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε υποχρέωση αναφορά, σε ποσοστώσεις, σε όρια και δεν έχουμε στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι ε, τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν θα είναι ποτέ αξιόπιστα. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε όσο το δυνατόν τεχνολογικά ουδέτεροι, αν θέλετε, και να μην προτείνουμε αυτήν ή την άλλη ε, τεχνολογική εναλλακτική λύση. Αλλά σίγουρα το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό. Γι' αυτό και προτείναμε και τα τηλέφωνα, τα smartphones. Υπάρχουν και άλλου είδους εξοπλισμοί. Υπάρχουν κάποια συστήματα, κουτιά, τα οποία σίγουρα δεν προϋποθέτουν καν την ε, παρέμβαση του Αλιέα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια συμμετοχή των ε, Αλιέων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας και βελτίωσης της ασφάλειας. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα σχόλια για το ότι επιβαρύνουμε του αλληλείς, ότι δεν είναι σε θέση πάντα να χρησιμοποιήσουν αυτό το τηλέφωνο και τον εξοπλισμό. Αλλά αυτό που ακούμε πολλές φορές από τους επιθεωρητές είναι ότι ναι, μπορεί να το κάνουν αυτό οι αλληλείς και το κάνουν όταν θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Όταν υπάρχει έλεγχος, ας πούμε, εκεί αμέσως ενημερώνουν και χρησιμοποιούν μια χαρά το τηλέφωνό τους. Εγώ αυτά ακούω. Επανέρχομαι σε αυτό που ήθελα να πω από την αρχή. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το ίδιο σύστημα για όλα τις κατηγορίες σκαφών. Υπάρχουν πολύ πιο απλά συστήματα για κάποιες κατηγορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να γενικευτούν. Ε, επαναλαμβάνω ότι επειδή θέλουμε να είμαστε πολύ ουδέτεροι όσον αφορά την ε, εγκατάσταση το θέμα της τεχνολογίας δεν είναι δική μας επιλογή. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να εγκατασταθούν ε, CCTV, όμως, δηλαδή τηλεοράσεις κυκλού, ε, κλειστού κυκλώματος. Όμως δεν επιβάλλουμε εμείς ποια τεχνολογία και ποια μάρκα. Λέμε απλώς ότι θα πρέπει να είναι συμβατή με τα δικά μας συστήματα. Δεν δίνουμε ιδιαίτερα στοιχεία όσον αφορά το πώς θα πρέπει να γίνεται η ανάλυση, αν θα γίνεται με το χέρι. Όλα αυτά μπορεί να τα επιλέξει. Ο καθένας θα πρέπει απλώς να είναι συστήματα συμβατά με αυτά που έχουμε και χρησιμοποιούμε. Και αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής. Όποια και να είναι η νομοθεσία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον, βεβαίως θα πρέπει να γίνονται σεβαστά όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ε, ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν ε, νομοθεσία για την ε, παρουσία κάμερας στον επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Αυτό ισχύει παραδείγματος χάρη στα σούπερ μάρκετ, στο δρόμο. Και όλοι αυτοί οι κανόνες ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν ε, παράδειγμα και σε άλλους χώρες. Πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο, λέει ο Πρόεδρος πρέπει δυστυχώς να σας ζητήσω να ολοκληρώσετε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, καταλαβαίνω ότι σημειώσετε πάρα πολλά, γιατί ακούσατε όλη αυτή τη συζήτηση. Όχι, ήθελα να σας πω και κάτι τελευταίο. Το θέμα της επιβολής ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συζήτησης. Αυτό δεν είναι κάτι το απόρριτο. Εννοείται ότι σήμερα δεν υλοποιείται η εφαρμογή ούτε οι κυρώσεις με ενιαίο τρόπο. Ε, in the ε, of 2020 a compliance. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση